Ladies and gentlemen, good morning. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Έχουμε πολλά πράγματα στην ημερήσια διάταξη και πολύ ενδιαφέροντα σήμερα, οπότε ας αρχίσουμε χωρίς καθυστέρηση. Επιτρέψτε μου πρώτα απ' όλα να σας ζητήσω να εγκρίνουμε την ημερήσια διάταξη για σήμερα και αύριο. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, θεωρείται εγκεκριμένη. Συμφωνεί. Καλώς. Τώρα στους φακέλους σας θα βρείτε και τα πρακτικά της προηγούμενης ε, συνεδριάσεω 11 και 12 Οκτωβρίου. Η προθεσμία για επιφυλάξεις, εφόσον έχετε παρατηρήσεις, προβληματισμούς, οτιδήποτε, είναι μέχρι το τέλος της συνεδρίασης αύριο. και της κοινή και της ε, δικιάς μας Επιτροπής Υποεπιτροπής ΣΕΝΤΕ. Αν δεν υπάρξουν παρατηρήσεις μέχρι τότε, τότε και τα πρακτικά θεωρούνται εγκεκριμένα. Δεν έχω ανακοινώσει της Προέδρου. Μια που, όπως είπαμε, Έχουμε πολλά θέματα στην ημερήσια διάταξη. Ας περάσουμε λοιπόν ευθύ αμέσω στο πρώτο ουσιαστικό σημείο της ημερήσιας διάταξης για σήμερα και είναι τα δίκτυα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της άμυνας και το μέλλον της αμυντικής έρευνας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με ιδιαίτερη χαρά λοιπόν, και θεωρώ ότι είναι προνόμιο για μένα, να υποδεχτώ εδώ τρεις εγκεκριμένους αναλυτές τους οποίους και θα σας παρουσιάσω κάπως σύντομα. Παρόλο που για πολλούς από εσά είναι γνωστοί και οι τρεις. Πρώτα απ' όλα έχουμε τον κύριο Κριστιαν Τεβιλμάνια, ο οποίος είναι διευθυντής του Γαλλογερμανικού Ινστιτούτου Ερευνών, Σαν Λουί, που είναι γνωστό το Ινστιτούτο αυτό, το Σαν Λουί. Και ο κύριος Βιλεμάνη θα μας το παρουσιάσει. Θα είναι ο πρώτος μας ομιλητής σήμερα. Στη συνέχεια θα ακούσουμε τον καθηγητή Πιότρο Σινκαρέτσικ, ο οποίος είναι Πολωνός, ακαδημαϊκός, διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Ερευνών αυτοματισμού και μετρήσεων στην ε, Βαρσοβία. Και μετά θα ακούσουμε τον τελευταίο μας ομιλητό για αυτό το θέμα, λόγω και λιγότερο σημαντικό βέβαια, τον κύριο Κλάου Τομά. Από ό,τι θυμάμαι, πάντα ήταν παρόν στα πάνελ μας, το θυμάμαι. είναι καθηγητής και ανώτερος σύμβουλος στο Ίδρυμα Φρανχόφερ στο Φράιμπουργκ. Φρανχόφερ λοιπόν, το Ινστιτούτο Φρανχόφερ. Οπότε κυρίες και κύριοι, η έρευνα στην άμυνα είναι κάτι ιδιαίτερο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπως θα θυμόμαστε, εδώ στο ΣΕΝΤΕ και με τον Κριστιαν ε, Λερ έχουμε συζητήσει και έχουμε πάρει αποφάσεις από αυτού. Μαζί με το Συμβούλιο. Οπότε θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον κύριο Βιλμάνια για να μας παρουσιάσει αυτό το θέμα. Έχετε το λόγο παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε για τα εισαγωγικά σας σχόλια. Μια που είμαι Γάλλος θα μου επιτρέψετε να μιλήσω γαλλικά. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι, όταν μιλάμε για την έρευνα και την τεχνολογία την αμυντική, δεν πρόκειται για έναν οποιοδήποτε τομέα εφαρμογή. Δουλεύουμε για άντρε και γυναίκε που θέτουν σε κίνδυνο την ίδια του τη ζωή και οι απειλές αυξάνονται. Εδώ στη διαφάνεια, αριστερά, να, το αποτέλεσμα της έκρηξης μιας ε, ελεγχόμενης ε, έκρηξης που κάναμε. Τα επόμενα χρόνια θα έχουμε και άλλες απειλές, εδώ τις βλέπετε, βαίνουν αυξανόμενες. Το Γαλλογερμανικό λοιπόν Ινστιτούτο Έρευνας αυτό το αντιλαμβάνεται. Αντιλαμβάνεται αυτή την ιδιαίτερη ευθύνη που έχουμε απέναντι στους ε, μαχημούς μας, ε, απέναντι στους στρατιώτες μας. Και έχουμε σαν στόχο πρώτα απ' όλα να προστατεύσουμε αυτούς τους μαχόμενους, αναπτύσσοντας τεχνολογίες ε, εντοπισμού των εχθρικών όπλων, αλλά και προκειμένου να αμβλύνουμε τις συνέπειες αυτών και να αναπτύξουμε και τεχνολογίες ε, προστασίας τους. Το δεύτερο που κάνουμε είναι να αναπτύσσουμε τεχνολογίες οι οποίες ε, στέλνουν στο στόχο την ε, κατάλληλη ενέργεια προκειμένου να δρανοποιήσουν τον εχθρικό στόχο, να τον καταστρέψουν και αυτό να γίνεται με χειρουργική ακρίβεια. Οι τεχνολογίες μας πρέπει να είναι ITAR free, το γνωρίζετε αυτόν τον ε, όρο, προκειμένου να ξέρουμε ότι η ζωή των ε, στρατιωτών μας μπορεί να μην έχει τιμή, έχει όμως ε, κόστος. Οπότε, συνεργαζόμαστε. Υπάρχουν χώρες που συμμετέχουν στο Ινστιτούτο μας και που δραστηριοποιούνται περισσότερο και άλλες που έχουν περισσότερο ένα ρόλο παρατηρητή. Η συνεργασία αυτή πάντω είναι ένα του, το οποίο θα μπορούσε κάλλιστα να διευρυνθεί και σε ολόκληρο το ευρωπαϊκό επίπεδο. Η πρακτική μα, η καθημερινή συνεργασία ε, χρησιμεύει ως καταλήτη σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας. Και αποφάσισα σήμερα να μοιραστώ μαζί σας κάποιες εμπειρίες που μας ε, διδάσκουν πώς να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της αμυντικής έρευνας και τεχνολογίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η έρευνα και η τεχνολογία από τον εμπορικό τομέα φυσικά είναι πολύ περισσότερο παρούσα σήμερα από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Αλλά υπάρχουν στρατιωτικές ιδιαιτερότητες και έτσι δύσκολα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ε, την τεχνολογία για μη στρατιωτικού σκοπού στο στρατιωτικό τομέα. Χρειάζεται μια παραπάνω προσπάθεια και έρευνα. Και θα σας δώσω ένα παράδειγμα, την ακουστική προστασία που είναι ένα μηχάνημα το οποίο αμβλύνει το θόρυβο. Αριστερά βλέπετε το μηχάνημα που χρησιμοποιείται στα αεροπλάνα και το οποίο μειώνει τον ε, θόρυβο. Δεξιά βλέπετε στην ίδια διαφάνεια την ε, ενεργό ακουστική προστασία που έχουμε αναπτύξει εμείς στο Ινστιτούτο μας ε, δηλαδή και που επιτρέπει στους στρατιώτες να ακούνε μεν τους ε, συναδέρφους τους, αλλά προστατεύεται το αυτί τους και δεν κινδυνεύουν τόσο πολύ από το φοβερό θόρυβο που μπορεί να κάνει ένα οστικό κύμα. Αυτό για να σας πω ότι οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται για μη στρατιωτικούς σκοπούς δεν μπορούν αυτές καθ' να χρησιμοποιηθούν και στο στρατιωτικό τομέα. Τώρα έχει μειωθεί ο προπολογισμό στην έρευνα και την τεχνολογία της ε, άμυνας και έχουμε και μεγάλη απώλεια ικανοτήτων δυστυχώς. Τα γνωρίζει αυτά βέβαια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προσπαθεί να προτείνει λύσεις. Και για να σας δώσω ένα παράδειγμα από το Ινστιτούτο μας, μας ζητήθηκε να ξαναχρησιμοποιήσουμε παλιότερη τεχνολογία, λεγόμενη munition flash, κάτι το οποίο όμως έχουμε καταλήψει κανονικά εδώ και πάρα πολύ καιρό. Χρειάζεται λοιπόν να κάνουμε νέε επενδύσει για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε την τεχνολογία. Συνήθω περνάμε από τρία στάδια. Συχνά λέμε ότι επιταχύνεται η τεχνολογία. Όμω αυτό είναι μερικό μόνο αλήθεια. Γιατί πρέπει να αναλύσουμε τι σημαίνει συνολικά η τεχνολογική πρόοδος. Αυτό το οποίο επιταχύνεται τελικά είναι η ανάπτυξη χρήσης των νέων τεχνολογιών. Όμως η ανάπτυξη αυτών των νέων τεχνολογιών χρειάζεται πάντα πάρα πολύ χρόνο. Πρέπει λοιπόν να συνοδεύσουμε αυτή την έρευνα όσο αυτή αναπτύσσεται. Εμείς ε, έχουμε χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα έρευνας ε, που μπορούμε και αυτό σε συνεργασία με άλλες χώρες, με χώρες του ΝΑΤΟ, σε συμβάσεις DARPA για παράδειγμα με τους Αμερικανούς ή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με τον ορίζοντα 2020, το ΠΑΝΤΡΑ ή τα συμβόλαια με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Εμείς πιστεύουμε λοιπόν ότι αυτά που έχουμε κάνει στη Γαλλία είναι πολύ πιο προηγμένα από ό,τι έχει γίνει οπουδήποτε αλλού όσον αφορά τα στάδια έρευνας. Χρησιμοποιούμε υποτροφίες για διπλωματικές εργασίες για παράδειγμα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πιστεύουμε ότι θα έπρεπε να εμπνευστεί από τέτοιε ιδέε και ίσω να χρησιμοποιήσει, να δημιουργήσει ένα κύτταρο τύπου DARPA ή Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνα χωρίς βέβαια να ξεχνάμε και την χρηματοδότηση των ορών, κάτι που είναι αναγκαίο για να διατηρηθεί η έρευνα και στο χρόνο. Το Ίδρυμά μας, που είναι γαλλογερμανικό όπως είπαμε, έχει μια μοναδική ιδιαιτερότητα μεταξύ άλλων ερευνητικών Ινστιτούτων Έρευνας και αυτή η ιδιαιτερότητα είναι ότι είναι διεθνές. Τι σημαίνει το να βάζουμε μαζί ερευνητές και μηχανικούς διαφορετικών υπηκοτήτων. Ξέρετε τον Οργανισμό Επιστήμης και Τεχνολογίας ε, του ΝΑΤΟ. Είναι ένα τεράστιο όργανο όπου όμως δεν συμμετέχουν μαζί στον ίδιο χώρο διαφορετική προέλευση ερευνητές. Έχει πάρα πολλούς ερευνητές, 5.000, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι προσφέρει λοιπόν αυτός ο οργανισμός επιτρέπει σε κάθε χώρα να αξιολογήσει την κατάσταση πραγμάτων όσον αφορά την τεχνολογία άμυνας. Να τοποθετηθεί σε σχέση με αυτή την κατάσταση, να ε, εκτιμήσει το βαθμό διαλειτουργικότητας και πολλές φορές και να επιτεχύνει και την, ε, τις επιλογές ε, τις τεχνολογικές που κάνει παρατηρώντας τι κάνουν οι διάφοροι εταίροι. Πολύ καλά είναι όλα αυτά, λένε περιορισμένα. Καλό θα ήταν να μπορούσαμε από κοινού να προχωρήσουμε σε καινοτομίες για την άμυνα που θα μας βοηθήσουν σε νέα προγράμματα. Το κάνει αυτό αυτός ο οργανισμός. Δεν το κάνει. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ή το κάνει σπάνια. Τα περισσότερα προγράμματα εξοπλισμών και συνεργασίας βασίζονται σε συμπράξεις όπου ο είναι στη χώρα του, στο κομματάκι του και είδαμε ότι αυτό δεν είναι αποτελεσματικό. Κάποιοι παλιότεροι λένε μάλιστα ότι προγράμματα συνεργασίας με νη εταίρους στοιχίζουν ρίζα νη φορές περισσότερο από ότι αν ε, είχαν ε, φτιαχτεί χωριστά από τον καθένα στη χώρα του. Εμείς λοιπόν μπορούμε να φροντίσουμε το ένα συν ένα να μην κάνουν δύο, αλλά παραπάνω από δύο. Αλλά αυτό μόνο αν μπορέσουμε αμοιβαία να προχωρήσουμε, να συνεργαστούμε δηλαδή και να νιώσουμε τις διαφορές μεταξύ μας σαν κάτι που πλουτίζει το έργο μας και όχι σαν εμπόδιο. Για να το πετύχουμε λοιπόν, η μόνη λύση είναι να βάζουμε ομάδες από διαφορετικές χώρες να συνεργαστούν μαζί. Δεν είναι επειδή βάζετε ένα like σε κάποιον στην άλλη άκρη του κόσμου που τον έχετε κάνει και φίλο σας. Αυτό δεν ισχύει. Γι' αυτό λοιπόν και θα πρέπει να προχωρήσουμε στην εξημέρωση, στην εξοικείωση. Και αυτό γίνεται μόνο με το συχνοτισμό, όπως έχει πει και στο μικρό πρίγκιπα ο Σαντεξουμπερί. Μόνο λοιπόν με αυτή την εμπειρία του να βρισκόμαστε μαζί στον ίδιο χώρο θα μπορέσουμε να αποκτήσουμε τέτοιες εμπειρίες από κοινού. Εμείς δουλεύουμε εδώ και 60 χρόνια και δουλεύουμε από κοινού διάφορες υπηκότητες μαζί και είναι αυτό που ζούμε ε, καθημερινά στο χώρο μας. Έχουμε 300 ε, μόνο ανθρώπους ε, που δουλεύουν, αλλά η ανταλλαγή εμπειριών είναι συνεχής. Και έτσι έχουμε και καλύτερη ποιότητα αποτελεσμάτων και αυτό το καταφέρνουμε παρόλο που έχουμε πολύ λίγους ακριβώς επειδή είμαστε από διαφορετικές προελεύσεις. Είμαστε πεπισμένοι δηλαδή ότι αυτός ο συγκνωτισμός, αυτή η συνύπαρξη επιστημόνων από διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους και από διαφορετικές χώρες αποτελεί και το κλειδί της επιτυχίας μας. Γι' αυτό και θα έπρεπε να επεκταθεί αυτό, αυτή η προσπάθεια, αυτό το πείραμα σε διάφορα κέντρα αριστείας όπου να χρησιμοποιούν επιστήμονες από διαφορετικούς κλάδους και από διαφορετικές ε, προελεύσεις. Όμως θα έπρεπε να γενικευθεί αυτό το πείραμα. Δεν θα ήταν ρεαλιστικό αυτό και ούτε καν αναγκαίο. Πρέπει όμως αυτό να γίνεται αρκετά ώστε να χρησιμεύσει ως καταλήτης προκειμένου το ένα συν ένα να μην κάνουν δύο αλλά πάνω από δύο. Στη χημεία ξέρουμε ότι ο καταλήτης είναι μια ουσία που χρησιμοποιείται σε μικρή ποσότητα προκειμένου να αυξήσει την ταχύτητα μιας αντίδρασης. Πώς γίνεται αυτό λοιπόν με 400 που είναι ο μέσος όρος ενό του Φρανχόβερ για παράδειγμα. Εμείς εποφελούμεθα από πολλά ακαδημαϊκά πανεπιστημιακά εργαστήρια με τα οποία μοιραζόμαστε τις ε, μεταπτυχιακές, ε, τις διπλωματικές εργασίες. Έχουμε δηλαδή διάφορους ε, υποψήφιους για ντοκτορά οι οποίοι δουλεύουν σε εμά. Και έτσι μοιραζόμαστε τη δουλειά που γίνεται στα πανεπιστημιακά εργαστήρια με το δικό μας Ινστιτούτο. Αυτό ακριβώς αποτελεί και τη μόχλευση και αυτή η μόχλευση είναι κάτι ζωτική σημασίας για μας και το αποτέλεσμα είναι όλοι να κερδίζουμε από αυτό και οι χώρες μέλη από τις οποίες προέρχεται ο φοιτητή γιατί παίρνουν πίσω έναν περισσότερο καταρτισμένο ε, επιστήμονα και εμεί βέβαια. Την προηγούμενη εβδομάδα ήμασταν στη Βιέννη, στην Αυστρία, για να προωθήσουμε ακριβώς ε, αυτό το μοντέλο στον ε, διευθυντή του ε, εθνικού των Εθνικών Εξοπλισμών και στην Επιστημονική Ακαδημία και υποδέχτηκαν τις ιδέες μας με ενθουσιασμό. Ένα λοιπόν τοκτορά το οποίο μοιραζόμαστε εμείς στο Ινστιτούτο μας και ένα ε, ακαδημαϊκό πανεπιστημιακό εργαστήριο που βρίσκεται κάπου αλλού, είτε είναι στην Πολωνία είτε οπουδήποτε αλλού, είναι κάτι πολύ θετικό. Είναι βέβαια και περίπλοκο γιατί για να διατηρήσει κανείς μια τέτοια σχέση αυτό κοστίζει. Τη λειτουργία αυτή θα πρέπει να την προωθήσουμε σε πανευρωπαϊκό επίπεδο μέσω ενός μηχανισμού που να αποτελεί το κίνητρο. Χρειαζόμαστε ένα απλό μοντέλο, όπου η μόνη δέσμευση για τους ε, οργανισμούς που συμμετέχουν είναι να ανταποκρίνονται σε μία χάρτα που πιστοποιεί την ποιότητα. Ένα απλό μοντέλο, το οποίο δεν θα βάζει ανταγωνισμό τον ένα με τον άλλον, αλλά όπου οι φοιτητέ θα επιλέγουν σε ποιο κέντρο αριστείας πιστοποιημένο ε, θέλουν να πάνε γιατί ανταποκρίνεται στη διπλωματική τους. Αυτό μπορεί να είναι το έρασμος. Φυσικά θα πρέπει να γίνουν προσαρμογές στον τομέα της ε, έρευνας και της τεχνολογίας στην άμυνα. Έτσι, φανταστείτε ένα έρασμος για την άμυνα. Ένα Ινστιτούτο λοιπόν έρευνας λειτουργεί όπως ε, το Ινστιτούτο μας, ε, βρίσκεται εδώ κοντά. Πρόκειται για το Von Carmen Institute, πραγματικά εδώ κοντά. Ε, εκεί πολλές χώρες συμμετέχουν σε συζητήσεις προκειμένου σταδιακά να καταρτήσουν περισσότερο κόσμο. Αυτά λοιπόν ε, είχα να σας πω σε λίγα λεπτά και για να συνοψίσω θα έρθω σε τρεις ε, συγκεκριμένες προτάσεις. για το επόμενο πρόγραμμα έρευνας και τεχνολογίας ε, για την άμυνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη στήριξη της έρευνας για την ε, άμυνα. Κάποια επιτόπου σχέδια και προγράμματα δεν φτάνουν. Δεύτερον, να προωθήσουμε και να στηρίξουμε τα κέντρα ε, αριστείας, τα πολυκλαδικά, με συμμετοχή πολλών χωρών. Και τρίτον, να προωθήσουμε και να στηρίξουμε ανταλλαγές μεταξύ επιστημόνων προς και από τα κέντρα αριστείας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε. Και τώρα το λόγο θα δώσουμε τον κύριο Πιότ Σινκάρτσικ, ο οποίος είναι ο διευθυντής του βιομηχανικού Ιδρύματος Έρευνας για Αυτοματοποίηση και Μετρήσεις της Βαρσοβίας. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη τιμή που ήρθα εδώ για να σας κάνω αυτή την παρουσία όσον αφορά τα μη επανδρομένα οχήματα. Ονομάζομαι Πίτερ Σινκάρτσικ και είμαι ο διευθυντής του ΠΙΑΠ ε, που είναι ένα ε, ίδρυμα ερευνητικό στην Βαρσοβία. Είμαστε ένα από τα δέκα κορυφαία τέτοια ιδρύματα στην Πολωνία. Έχουν προσταμένη αρχή το Υπουργείο ανάπτυξη και μέχρι σήμερα είμαστε οι μόνοι που παράγουν αυτά τα ειδικά ρομπότ ε, που χρησιμοποιούν διάφορε εφαρμογέ και συγκεκριμένα αυτά τα ρομπότ χρησιμοποιούνται στην ε, έρευνα και στην άμυνα. Αυτοματοποίηση και χρήση ρομπότ για την ε, παραγωγή, για τη γραμμή παραγωγής και χρησιμοποιούνται επίσης από την αστυνομία, το στρατό και άλλες ε, υπηρεσίες ε, πολιτικής προστασίας. Επίσης, ε, διεξάγουμε έρευνα βιομηχανικού χαρακτήρα και διάφορες άλλες βιομηχανικές εφαρμογές και επίσης οργανώνουμε το οτομάτικον που είναι η μεγαλύτερη έκθεση Ανατολικής Ευρώπης και επίσης διάφορες άλλες διασκέψεις επιστημονικές ε, επιμελούμεθα την έκδοση διαφόρων ε, περιοδικών εκδόσεων ε, που ενδιαφέρουν μηχανικούς, επιστήμονες. Επίσης εκπαιδεύουμε στον τομέα της βιομηχανίας εργαστήρια, σεμινάρια, διάφορες συναφείς εκδηλώσεις οργανώνουμε και κάθε χρόνο μας απονέμουν 30 με 50 διεθνή βραβεία. Επίσης, έχουμε και 30 έως 50 τεχνίες, οι οποίες κατοχυρώνουμε κάθε χρόνο. Από το 1991 ξεκίνησε η διεθνής μας συνεργασία. Επρόκειτο για το πρόγραμμα πλαίσιο υπαριθμών 3 και έχουμε περίπου 100 διεθνή προγράμματα και 10 εξ αυτών των προγραμμάτων έχουν εμάς ως συντονιστές. Και το τάλος ήταν ένα από τα μεγαλύτερα εξόδων των προγραμμάτων. Χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του πρώτου πλαίσιου προθυμών 7, 20 εκατομμύρια ευρώ και επίση υπήρξε συντονισμό ενό μεγάλου επιχειρηματικού κονσότσιουμ και είχαμε από παντού, από Ευρώπη και Ισραήλ, διάφορους ε, που συμμετέσχουν. Ο σκοπός ήταν να έχουμε κάποιο είδους ανάπτυξη συστήματος φύλαξης των Ευρωπαϊκών Συνόρων με την χρήση μη επανδρομένων ε, οχημάτων εδάφους. Τα, θα, τα λέμε UGV. Έχουμε δύο είδη ε, τέτοιων οχημάτων. Το ένα για την φύλαξη των συνόρων και επισήμανση ε, εισβολέων με κάποιους αισθητήρε και επίσης είχαμε ένα άλλο UGV ε, το οποίο μπορεί να τους πιάσει, να τους συλλάβει αυτούς τους εισβολείς. Οπότε και θέσαμε σε εμπορία αυτά τα αποτελέσματα της επιστημονικής μας έρευνας. Οπότε και ξεκίνησε το πρόγραμμα Eden, στα πλαίσια του οποίου αναπτύξαμε κάποιους αισθητήρε, κάποια εργαλεία για την αντιμετώπιση κάποιων απειλών ε, που έχουν σχέση με εκρηκτικά, με χημικά όπλα και με κυβερνοεπιθέσεις. Για να δούμε τώρα τι άλλες δραστηριότητες έχουμε. έχουμε διάφορα προγράμματα στα πλαίσια του ορίζοντα του 2020, μην πω στις λεπτομέρειες τώρα, αλλά πάντως έχουμε έρθει σε επαφή και συνεργασία με πολλές άλλες υπηρεσίες ε, αμυντικών υπηρεσιών, όπως το Μούσας, οπότε έχουμε και αυτή την κινητή πλατφόρμα για να ανοιχνεύονται στις πολεμικές ζώνες οι ελεύθεροι σκοπευτές. Επίση, κάνουμε και κάποιες μελέτες σκοπιμότητας και διάφορους χάρτες ε, σε σχέση πάντα με, τι με τις εφαρμογές των ε, ε, μη επανδρομένων οχημάτων. Τώρα σε αυτή τη διαφάνεια μπορείτε να δείτε διάφορα ρομπότ τα οποία παράγουμε και τα οποία θέτουμε σε εμπορία και τα πουλάμε σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως και χρησιμοποιούνται και στην Πολωνία, αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, στη Μέση Ανατολή, αλλά και στην Αφρική. Όμω δεν σταματάει εκεί η παραγωγή των ρομπότ από πλευρά μα για του πελάτε μα, Έχουμε και άλλα ρομπότ τα οποία δεν απεικονίζονται εδώ. Για να πούμε τώρα δύο λόγια όσον αφορά αυτά τα UGVs, δηλαδή τα, μη πανδρομένα οχήματα εδάφους. Ο βασικό σκοπό είναι να προστατεύουν το προσωπικό από τις απειλές Βλέπετε εδώ αριστερά, πάνω πάνω βλέπετε ε, ε, κάποιον ο οποίος ασχολείται με κάποια βόμβα, να μια απειλή που μπορεί να προερχέται από την ύπαρξη, την ενδεχόμενη κάποιων εκρηκτικών. Και δεξιά βλέπετε ότι το πρόσωπο αυτό που ασχολείται με το κριτικό είναι ασφαλή. Τώρα τι κάνουμε με αυτά τα ε, οχήματα. Πρώτα πρώτα έχουμε την εναρκαλίευση και κατόπιν έχουμε άλλους ελέγχους που διεξάγονται και σε χώρους ε, ε, μη στρατιωτικούς, φύλαξη, περιπολία. Δεξιά βλέπετε το όχημα που κάνει αυτή την περιπολία και μετά έχετε και άλλα ρομπότ που εδώ στις εικόνες σας που δεν είναι κινούμενα αλλά για κοιτάξτε το καλύτερα. Εδώ αριστερά μπορεί να δείτε ένα άλλο ρομπότ. Κορεατικό. Αυτό ασχολείται με την φύλαξη συνόρων μεταξύ Βορείων Νοτιο και βλέπετε πέρα να υπάρχει ένα πολυβόλο για ένας υπολογιστής οπότε μπορεί να πυροβολήσει τους ε, εισβολείς με δική του πρωτοβουλία χωρίς να λάβει εντολή από άνθρωπο. Βέβαια εδώ πέρα υπάρχουν διάφορα ηθικά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη όσον αφορά το τρέξιμο, την εκτέλεση προγράμματος. Ε, μετά βλέπετε κάποια άλλα τα οποία αφορούν την ε, κένωση κάποιων τραυματισμένων από την ε, επικίνδυνη ζώνη. Επίσης ε, βλέπετε άλλα ρομπότ για άλλους ελέγχους ε, και βιομηχανικών χρήσεων ένα άλλο για αντιμετώπιση πυρκαγιών, επίσης τα άλλα που ασχολούνται με εκρηκτικά και την εξοδετέρωσή τους. Στην επόμενη διαφάνεια βλέπετε άλλα παραδείγματα ε, χρήσεων διαφόρων ρομπότ που παράγουμε. Εδώ βλέπετε κάποιες άλλες εφαρμογές τεχνητικού χαρακτήρα, επιμελητία για τον στρατό, ε, τα οποία παράγονται από το Ίδρυμά μας στην Βαρσοβία και δεξιά μια κλασική εφαρμογή εκεί που το ρομπότ κουβαλάει το, το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί από τον στρατιώτη. Επίσης χρησιμοποιούνται άλλα ρομπότ και από σταθμούς παραγωγής ενεργείας ε, άλλα έχουν ζωμηθεί στην Φουκουσίμα και άλλες εφαρμογές αφορούν ε, σεισμοπαθείς και ατυχήματα σε κατασκευές, σε οικοδομές και έχουν χρησιμοποιηθεί ρομπότ δικά μας και στα τραγικά γεγονότα που ε, συνέβησαν στο World Trade Center της Αμερικής. Ίσως θυμάστε ότι έχουμε ξανασυζητήσει για τα αυτόνομα συστήματα ε, που φέρουν όπλα και αυτά είναι δηλαδή κάποια οχήματα και πολλές χώρες προσπαθούν να βρουν λύσεις στα σχετικά προβλήματα εκτός από μας Έχουμε επιστήμονες που ασχολούνται με αυτά τα ρομπότ και υπάρχει δραστηριότητα ευξημένη και έντονη και στη Ρωσία για το ίδιο θέμα. και αυτά τα εξοπλισμένα, τα ένοπλα, στα πούμε, οχήματα και ρομπότ έχουν χρησιμοποιηθεί σε πραγματικές συνθήκες πολεμικές, όπως την ε, Συρία και η χρήση τους ήταν επιτυχής. Τώρα κάποιες προτάσεις και συστάσεις μας. Τι θα πρέπει να μελετηθεί, να ληφθεί υπόψη από τη δική μας οπτική γωνία όσον αφορά τα δικά μας θέματα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να σκεφτούμε το να ξεκινήσει κάποιο διεθνές πρόγραμμα το οποίο να έχει σχέση με τον σχεδιασμό τέτοιων ε, μη επανδρομένων οχημάτων στην Ευρώπη και να φτιάξουμε κάποιες πλατφόρμες, λέω πλατφόρμες πολλές και όχι μία, γιατί δεν υπάρχει μία λύση για όλες τις εφαρμογές. βέβαια να υπάρχει διαλειτουργικότητα μεταξύ των διαφορετικών εργαλείων και αισθητήρων. Ε, να επιδέχεται το σύστημα αυτό ε, τον συνδυασμό και να υπάρχει συνεργασία μεταξύ των ρομπότ. Και μπορεί το ένα ρομπότ να βοηθά το άλλο όταν υπάρχει θέμα δράσης σε πολεμική ζώνη. Ε, επίσης, θα πρέπει να υπάρχει ισορροπία όσον αφορά τη βιομηχανία και την ε, έρευνα και επίσης ισορροπία από γεωγραφική σκοπιάς. Αυτό το μοντέλο έχει χρησιμοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος. Όταν η Πολωνία προσχώρησε στην υπηρεσία διαστήματος. Ξεκίνησε το πρόγραμμα αυτό και ο σκοπός ήταν να βοηθηθεί η Πολωνία που μόλις είχε προσχωρήσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ούτως ώστε ε, να μπορεί να κινηθεί στην αγορά του διαστήματος με ίσους όρους όπως η, τα παλαιότερα μέλη. υπάρχουν κάποιες ενισχύσεις όσον αφορά το know-how, όσον αφορά την κατάρτιση και υπάρχει μια εποπτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων. Εδώ θα, θα βάλω τελεία και θα σας ευχαριστήσω για την προσοχή σας. Εμείς ευχαριστούμε κύριε καθηγητά. Και τώρα ο καθηγητής Κλάους Τόμα που προέρχεται από την εταιρεία το φορέα Φράνχοφερ του Φράιμπουργκ. Θα μιλήσω και εγώ γερμανικά. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαίρομαι πάρα πολύ που μπορώ να σας παρουσιάσω τις ιδέες μου ε, και τα θέματα της αμυντικής έρευνας. Από που προέρχομαι από τον όμιλο Fraunhofer ε, για εφαρμοσμένη έρευνα είναι από τους μεγαλύτερους ομίλους στην Ευρώπη ολόκληρη και στη Γερμανία. 24.000 υπαλλήλους έχουμε 69 Ινστιτούτα σε όλη τη Γερμανία, το βλέπετε από το χάρτη, 2,1 δις ο συνολικός προϋπολογισμός μας. 70% του προϋπολογισμού πρέπει να τα κερδίζουμε εμείς από πληρωμένη έρευνα, από την βιομηχανία κυρίως, αλλά και από δημόσιους φορείς και από κυβερνήσεις. Ποιους τομείς καλύπτουμε θα τους βρείτε στην επόμενη διαφάνεια. Ε, έχουμε κατανείμει σε διάφορες ομάδες την έρευνα που κάνουμε, ε, καινοτομία, τέσσερα Ινστιτούτα έχουν συνδεθεί για να κάνουν έρευνα για το μέλλον. Έχουμε πολύ μεγάλο όμιλο που ασχολείται με τεχνολογίες πληροφορίας, κυβερνοτεχνολογία. Έχουμε βιολογικές επιστήμες, βιολογία και ιατρική τεχνολογία. Έχουμε μια ομάδα που ασχολείται με την ε, οπτική και ηλεκτρονική και τα λέιζερ. Έχουμε τεράστιο τμήμα που αφορά τη μικροηλεκτρονική αυτή τη στιγμή και φυσικά έχουμε και τεχνική παραγωγής και που εδρεύουν όλα αυτά στο Στουτκάρδη, στο Άχεν. Ε, έχουμε μια ιδιαιτερότητα, έχουμε ξεχωριστό τομέα 10 Ινστιτούτων που ασχολούνται με την ε, έρευνα για την ε, ασφάλεια και την άμυνα. Το 2022 συστήθηκε. Τι θέλω να συζητήσω μαζί σας. Έχουμε κάνει ήδη σημαντικά βήματα για μια επιτυχή στρατηγική ε, να στηθεί αμυντική έρευνα στην Ευρώπη. Αυτό άρχισε με μια συνολική και παγκόσμια στρατηγική ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχει σημαντικούς στόχους. Και παράλληλα με αυτή την Global Strategy έχει συσταθεί και μια ομάδα προσωπικότητων που έχει σημαντικές ιδέες και θα ήθελα λίγο να αναφερθώ σε αυτή. Αμέσως μετά ε, ήρθε το πολιτικό πρόγραμμα για την αμυντική έρευνα. Αυτά τα γνωρίζετε εσείς και εσείς τα επιβάλλετε μάλιστα. Ήταν ορόσημο πραγματικό αυτό ε, το γεγονός ότι καταφέρατε για πρώτη φορά να το επιβάλλετε, για πρώτη φορά να χρηματοδοτείτε αμυντική έρευνα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα ε, υπάρχει και μια άλλη διαδικασία, το πρόγραμμα δράσης για την άμυνα. Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος δράσης έχουμε τώρα την προπαρασκευαστική δράση που ξεκίνησε φέτος και η οποία ε, θα αποτελέσει ουσιαστικά τη βάση για μια ε, μεγαλύτερη προσπάθεια ενός ερευνητικού προγράμματος πανευρωπαϊκού. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω ένα πλαίσιο ε, με τέσσερις πυλώνες, έτσι το έχω ονομάσει, για το πώς θα μπορούσε να προχωρήσει η έρευνα στα θέματα της αμυντικής βιομηχανίας. Θυμίζονται ένα σημαντικό έγγραφο, τη συνολική στρατηγική, όπου ορίζεται πραγματικά ο φιλόδοξος στόχος και τα φιλόδοξα σχέδια που έχουμε για την Ευρώπη, πώς θέλουμε παγκοσμίω να εγγραφεί η Ευρώπη, είναι ένα κομβικό έγγραφο, απορρέουν πολλά από αυτό. Ήδη σας ανέφερα προηγουμένως ότι παράλληλα ε, με την παγκόσμια στρατηγική έχουμε εργασίες ε, της ομάδας προσωπικότητων. Βλέπετε εδώ μερικές προσωπικότητες με την Επίτροπο Μπιενκόφσκα στο κέντρο, στην οποία επιδώσαμε στις 23 Φλεβάριου του 2016 την έκθεση Βλέπετε και τον επικεφαλής της ΕΝΤΑ, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας ε, και τον ε, πρόεδρο του Fraunhofer Institute, τον ε, προϊστάμενό μου και άλλες προσωπικότητες από τη βιομηχανία. Ποια είναι τα βασικά που προτείνουν αυτοί αυτές οι προσωπικότητες, να χρησιμοποιηθεί η αμυντική συνεργασία για την έρευνα, έτσι ώστε η Ευρώπη να είναι ένας πάροχος ασφαλείας, ένας εγγυητής σε θέματα ασφαλείας και αξιόπιστος εταίρος σε ένα παγκόσμιο επίπεδο. Προτείνουμε επίσης η Ευρωπαϊκή Αμυντική Ερευνά να χρησιμοποιηθεί έτσι ώστε να σφυριλατηθούν συνεργασίες σε ελεγόμενες ε, τεχνολογίες κλειδιά και έτσι ώστε να χρησιμοποιηθούν και να δημιουργηθούν ικανότητες ε, για τις ευρωπαϊκές χώρες. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο το οποίο ακούσαμε και προηγουμένως θα πρέπει να σκεφτούμε τους ενεχομένους φορείς. Ε, περί τίνος πρόκειται εδώ βεβαίως κυβερνήσεις με μονομένες χώρες, Υπουργεία Άμυνας, ε, επίσης οι αμυντικές ε, βιομηχανίες που οπωσδήποτε τις χρειαζόμαστε και ε, ε, οι οργανισμοί έρευνας και τεχνολογίας που παρακάθονται και σήμερα εδώ. Όλους αυτούς τους φορείς θα πρέπει να τους ενώσουμε για να μπορεί η Ευρώπη να σταθεί στα πόδια της στα θέματα αυτά της έρευνας. Και πολύ σημαντικό που το λέει εδώ η τελευταία παράγραφος και το ακούσαμε και προηγουμένω, στρατηγική αυτονομία θα πρέπει να διαθέτει η Ευρώπη. Να το κοιτάξουμε πολύ προσεκτικά. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για να έχουμε μια τέτοια στρατηγική αυτονομία ή να τη διανοηθούμε καν, χρειαζόμαστε μια πολύ καλή τεχνολογική και βιομηχανική βάση σε θέματα αμυντικής τεχνολογίας. Στην επόμενη διαφάνεια προσπάθησα ε, να τα εξηγήσω όλα αυτά. Ποιοι είναι οι στόχοι, οι μεγάλη επίβολοι που έχουμε θέσει στην Ευρώπη. Οπωσδήποτε το θέμα ε, ε, τη μη εξάρτηση, αυτονομία, έστω και μερική της Ευρώπης. Οι κρίσιμες τεχνολογίες θα πρέπει να παράγονται στην Ευρώπη, θα πρέπει να τις έχουμε εδώ. Η αλυσίδα παραγωγής και supply chain θα πρέπει να είναι στην Ευρώπη χωρίς να χρειάζεται να εξαρτώμαστε από την Κίνα ή τις ΗΠΑ για σημαντικά στοιχεία αυτής της αλυσίδας. Για να γίνει αυτό χρειάζεται μια πολύ στιβαρή βιομηχανική βάση που θα πρέπει να είναι αηφόρα, βιώσιμη, διασυνδεδεμένη και φυσικά ανταγωνιστική. Άλλο σημαντικό σημείο για να ενισχυθεί η συνεργασία στην Ευρώπη, η αμυντική συνεργασία, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο το πρόγραμμα έρευνας, το ερευνητικό πρόγραμμα όπως έχουμε κάνει και στην πολιτική έρευνα όχι στη στρατιωτική και βεβαίως θα πρέπει να αυξήσουμε την αντίσταση της Ευρώπης και την αντοχή της σε μια παγκοσμιοποιημένη σημερινή πραγματικότητα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό για να αντέχει η Ευρώπη. Τούτων όλων λεχθέντων θα ήθελα να σας προτείνω σύντομα τι θα μπορούσαμε να κάνουμε ως βάση για τη συζήτηση και πλαίσιο έρευνας, τις τέσσερις πυλώνες που σας είπα και προηγουμένως, έτσι το έχω διαρθρώσει, να σας παρουσιάσω ε, τους τέσσερις πυλώνες αυτούς επιγραμματικά. Πρώτο, θα πρέπει να πάρουμε αυτή τη στρατηγική οδό για να ενισχύσουμε τις δυνατότητες. Ο, ο αμυντικός οργανισμός έχει δει μια προσπάθεια, θα πρέπει να τη διευρύνουμε και αυτή τη στιγμή ορίσουμε ποιε είναι οι στρατιωτικέ και αμυντικέ δυνατότητες Ευρώπης ανάλογα να προσαρμόσουμε και τα ερευνητικά μας προγράμματα. Αυτά ε, σε βιομηχανικό επίπεδο. Αν σκεφτούμε όμως ε, τη πιο εφαρμοσμένη έρευνα, ε, παραμένει ένα ζήτημα αυτό των τεχνολογιών. Ποιε είναι οι βασικές τεχνολογίε κλειδιά που χρειαζόμαστε στην άμυνα. Άλλο πολύ σημαντικό είναι να δημιουργήσουμε ε, ευρωπαϊκά κλάστερ, όχι μόνο στην έρευνα, και στην έρευνα, αλλά και στην ανάπτυξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στη βιομηχανία και σε άλλες εταιρείες. Οι μικρομεσαίες ε, που ε, αναπτύσσουν σημαντικά προϊόντα ή τα παράγουν κιόλας. Και ένα πολύ σημαντικό, το τέταρτο είναι αυτό που χρειαζόμαστε, ένα φόρουμ, ένα δίκτυο ε, θεσμών που να κάνουν το στρατηγικό σχεδιασμό και να έχουν μια προοπτική 30 ετών σε βάθος χρόνου και μας κάνουν προτάσεις ε, για τις ανάγκες τους. Τώρα, να μπω ε, στους διάφορους πυλώνες πιο λεπτομεριακά. Για τον πρώτο πυλώνα, θα πρέπει να ορίσουμε πραγματικά τι εστί defense capability. Κάθε κράτος έχει τη δική του ε, πολιτική, το δικό του σχεδιασμό, ανάλυση, τι χρειαζόμαστε, Γαλλία, ε, Γερμανία και για την Ευρώπη μπορεί να έχουμε ενιαίες ανάγκες. Ε, αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ποιε είναι αυτέ οι ικανότητε. Θα πρέπει στη συνέχεια να αναπτύξουμε κάποια ερευνητικά προγράμματα έτσι ώστε να καταλήξουμε σε κάποια προϊόντα, πρωτότυπα επίδειξη. αυτό αφορά τη βιομηχανία. Όταν ξέρουμε ποιε είναι οι ανάγκε μα. Στην επόμενη διαφάνεια, όταν ξεκίνησαν όλα, δεν ξέραμε τι θέλαμε ακριβώς, αλλά είπαμε ότι χρειαζόμαστε μια στρατηγική παγκόσμια ε, και μέσα σε αυτή τη στρατηγική θα υπάρχει ένα υποσύνολο που θα λέγεται αμυντική στρατηγική. Ε, θα πρέπει να καθορίσουμε ποιες ικανότητες θέλουμε να έχει η Ευρώπη, ευρωπαϊκές αποστολές ε, στην άμυνα και στη συνέχεια να δούμε πώς θα συνενωθούμε, πώς θα συνεργαστούμε για να το επιβάλλουμε Γι' αυτό χρειαζόμαστε ερευνητικό πρόγραμμα και αναπτυξιακό πρόγραμμα και στη συνέχεια προγράμματα για κοινέ προμήθειες. Δεύτερος πυλώνας. Μπαίνουμε τώρα στη θεμελιώδη έρευνα θα πρέπει να βρούμε ποιες είναι οι βασικές αμυντικές τεχνολογίες, key defense technologies. Ξέρετε ότι και στην πολιτική έρευνα υπάρχουν κάποια όργανα που συνεδριάζουν παγίως και ε, βλέπουν ποιες είναι οι βασικές τεχνολογίες που χρειάζονται και που πρέπει να γίνει έρευνα. Τα ίδια ισχύουν και για την άμυνα. Υπάρχουν στρατηγικές τεχνολογίες, καινοτομία, ε, αναδυόμενες τεχνολογίες, επαναστατικές τεχνολογίες. Ο καθένας λέει με διάφορα ονόματα. Πάντως ε, αυτό που χρειάζεται είναι οι βασικές τεχνολογίες να είναι διαθέσιμες για τα βιομηχανικά μας προγράμματα. Επιτρέψτε μου εδώ εμβόλυμα να πω κάτι. Ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο ε, που προέκυψε και από τη συζήτηση και εκ των Θα πρέπει οπωσδήποτε να πούμε ότι αυτό που μας νοιάζει δεν είναι να μοιράζουμε λεφτά στην Ευρώπη, να πάρουν διάφορα Ινστιτούτα και διάφορες εταιρείες. Όχι, θα πρέπει να έχουμε αποδεδειγμένη επιστημονική αριστεία και να αποδείξεις ότι έχεις το τεχνολογικό υπόβαθρο. Όχι να στήσουμε νέες δομές, αλλά όποιοι έχουν την εμπειρία και αποδεδειγμένα είναι επιτυχημένοι και έχουν κάποια πραγματογνωμοσύνη ε, να ε, λάβουν τη χρηματοδότηση. Το επόμενο δεν θα το σχολιάσω, μπορείτε να το διαβάσετε μόνοι σας, έχει λεπτομέρειες αυτή η διαφάνεια. Πάμε στον τρίτο πυλώνα, πολύ σημαντικό, τα ευρωπαϊκά κλάστερα αριστείας. Και εδώ δεν αναφέρομαι μόνο στην έρευνα, αλλά και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τεχνολογικά κέντρα, Ινστιτούτα στην Ευρώπη, να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο που είναι πάρα πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε. Έχουν ήδη ξεκινήσει κάποια πράγματα, μπορείτε να τη διαβάσετε σε αυτή τη διαφάνεια και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάποιες σκέψεις κάνει και κάποιες προτάσεις για να αναπτυχθεί ένα ευρωπαϊκό ε, δίκτυο περιφερειών που έχουν σχέση με την άμυνα. Βλέπετε το χάρτη τον ευρωπαϊκό εδώ και κάτω το link που υπάρχουν περιφέρειες δηλαδή όπου αναπτύσσεται αμυντική τεχνολογία και συγκεντρώνεται εκεί δεν είναι καθόλου πλήρης ο χάρτης αυτός, απλώς δείτε το παρακαλώ ως μια βάση για να καταλάβουμε τι χρειάζεται στην Ευρώπη, ποιες κυβερνήσεις ενέχονται, ποιες ε, περιφέρειες και να αρχίσουν να ε, διασυνδέονται μεταξύ τους οι μικρομεσές. Αυτό είναι χήμερα, τώρα είναι ρεαλιστικό. Καθόλου χήμερα δεν είναι. Ε, έχουμε και εμπειρία προηγούμενη. Εδώ και 10 χρόνια κάνουμε έρευνα σε θέματα ασφαλείας. Σας ε, δίνω ένα παράδειγμα τυχαίο, χαρακτηριστικό όμως, για την πολιτική έρευνα ασφαλείας. Ένα σχέδιο ολοκλήρωσης μεγάλη κλίμακα με 20 εταίρους από 10 ευρωπαϊκά κράτη, οι οποίοι συνενώθηκαν στην προσπάθεια αυτή, έτσι ώστε να αναπτύξουν μια συγκεκριμένη τεχνολογία ας πούμε, για σωστικά συνεργεία, για διάσωση τραυματιών σε περίπτωση θεομηνιών, για την πολιτική προστασία. Αυτό το δίκτυο θεσμών λειτουργεί, είναι ζωντανό, υπάρχουν πολλά έργα, πολλά σχέδια όπου συνδεδεμένα ε, συνεργάζονται και όποιος έχει μια ιδέα τηλεφωνεί στους συνεργάτες στην Ευρώπη και στους εταίρους και ε, πιστεύουμε ε, και θέλουμε να γίνει κάτι τέτοιο και στην άμυνα. Και τελευταίος πυλώνας είναι κάτι που χρειάζεται οπωσδήποτε ένα ευρωπαϊκό δίκτυο για το στρατηγικό σχεδιασμό και την ε, έρευνα στο μέλλον. Θα πρέπει να σκανάρουμε τον ορίζοντα, ας πούμε, foresight studies, παγκοσμίω να κοιτάξουμε υπάρχει τίποτα εκεί, έχει βγει καμιά νέα ιδέα για νέες τεχνολογίες, θα μπορούσε να μας ενδιαφέρει, να έχει σημασία για μας. Μια μόνιμη παρατήρηση της τεχνολογίας, τι προκύπτει, τι βγαίνει καινούριο, πώς μπορούμε να το αξιοποιήσουμε και πώς να το χρησιμοποιήσουμε στην ευρωπαϊκή αμυντική έρευνα. Θα πρέπει να βλέπουμε και ποιες είναι οι γεωπολιτικές τάσεις. Δεν χρειάζεται να σας τα εξηγήσω, τα κάνετε και εσείς στο Κοινοβούλιο. Ας πούμε, διαφαίνονται νέες απειλές, έχει αλλάξει ε, κάτι στις απειλές, ε, έγκαιρη προειδοποίηση. Μήπως υπάρχουν πουθενά νέε τεχνολογικές εξελίξεις που μας έχουν διαφύγει και μπορεί να έχουν σημασία για την άμυνα ή και επιπτώσεις στην άμυνα και την ασφάλειά μας. Αυτά. Τελευταία διαφάνεια. Σε ευχαριστώ που με ακούσατε και με χαρά ε, θα σας απαντήσω στη συζήτηση. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ όλους τους καθηγητές. Τώρα ερωτήσεις, απαντήσεις. Ο κύριος... Για τον κύριο να λυπάμαι για αυτό που έγινε με τη διερμηνία. Δεν υπάρχει διερμηνία στα τσεχικά. Μπορείτε όμως να μιλήσετε τσεχικά. Και θα μεταφραστούν τα τσεχικά. υπήρξε κάποιο πρόβλημα με την τσεχική καμπίνα, κάτι έκτακτο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Έλερ πρώτα. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα μιλήσω και εγώ γερμανικά. Θα ήθελα καταρχάς να πω το εξής. Χαιρόμαστε και για την παρουσία των μεγάλων Ινστιτούτων, ερευνητικών ιδρυμάτων και τη θετική απήχηση που είχε η πρωτοβουλία μας, πόσο την αγκάλιασαν. Εργάστηκε εδώ πολύ σκληρά και ο Μίχαελ Γκάλερ και πολλοί άλλοι χρόνια ολόκληρα πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Όχι μόνο για τον προϋπολογισμό, αλλά και για την πολιτική βούληση να ασχοληθούμε με αυτά τα θέματα. Έχω μια ερώτηση που μπορεί να είναι λίγο στενάχωρη, δεν είναι τόσο ευχάριστη. Ε, και προς τα οποία που το γνωρίζουμε από τα πολιτικά ερευνητικά προγράμματα. Μιλήσαμε πάρα πολύ για την έρευνα, για τις δομές. Σε αντίθετη με τα πολιτικά προγράμματα ασφαλείας, όπου στις προμήθειες έχουμε διάφορες αγορές, το, έχουμε ε, τον ιδιωτικό τομέα, έχουμε το δημόσιο ως πελάτες. Ε, ας πούμε, τίθεται το εξή ερώτημα. Για τις προμήθειες, λοιπόν, οι αγορές είναι εθνικές ε, για τις κρατικές προμήθειες ακόμα και εθνικές είναι και οι πολιτικές καταστάσεις κάθε φορά και τα δεδομένα. Ερωτώ, λοιπόν, το εξής η Πολωνία, η Τσεχία, η Ουγγαρία συνεχίζουν να ε, θεωρούν με επιφύλαξη κατά πόσο χρειάζεται μια ευρωπαϊκή πολιτική κοινή άμυνας και ασφάλειας. Είναι, ε, ε, τώρα ευκαιρία υπάρχει δυνατότητα να συνεργαστεί η έρευνα για να απορροφήσει τους απαραίτητους πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει προθυμία από τα κράτη αυτά πέρα από την έρευνα να συνεργαστούμε σε ένα κοινό πλαίσιο με κοινού στόχου, είτε είναι στρατηγική, είτε είναι τεχνολογική, αλλά στο κάτω-κάτω και μια κοινή ε, ευρωπαϊκή δομή για τις προμήθειες αμυντικού υλικού. Γιατί υπάρχει μια αντίφαση ότι τεχνολογικά υπάρχουν αυτά τα προγράμματα, αλλά αυτός δεν είναι ο απότερο στόχος. Ο απότερος στόχος είναι πολιτικός, δηλαδή μια κοινή ε, αμυντική ικανότητα της Ευρώπης και κοινή δυνατότητα ε, άρθρωσης αυτών των δυνατοτήτων και προβολής. Δηλαδή εσείς πώς το βλέπετε αυτό, την εθνική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Να συνεργαστούμε θέλουνε μόνο στην έρευνα ή μήπω και στην άμυνα. Για να έχουμε κοινού στόχους. Γιατί αυτό θα ήταν βασική προπόθεση. Αυτή ήταν η πρώτη μου ερώτηση. Ερώτηση δεύτερη. Προς όλους. Θέτουμε ευρωπαϊκούς στόχους εμείς, αλλά η σημαντική πραγματικότητα είναι εθνική ε, στην κάθε χώρα. Υπάρχουν κάποιες δομές ε, οι οποίες αποδίδουν και έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, αλλά αυτές είναι διμερείς διακυβερνητικές συνεργασίες. Εμείς υπάρχουν διάφορες δομές, καμιά σειρά στα διάφορα κράτη, διμερείς συνεργασίες. Εμείς ερχόμαστε να τις ανταγωνιστούμε αυτές τώρα. Ποια είναι η σχέση μας και σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε διμερές υπάρχουν κάποιες δομές και υπάρχουν και μεγάλα προβλήματα χρηματοδότησης. Και αυτά τα προβλήματα, τις τρύπες χρηματοδότησης θα τις βουλώσουμε τώρα με ευρωπαϊκά κονδύλια κατά κάποιο τρόπο. Αλλά όταν λέμε ότι έχουμε ένα κοινό ευρωπαϊκό στόχο, το ερώτημα είναι αυτή η εμπειρία πώς αξιοποιείται που είναι διμερής. Είναι ρεαλιστικό τώρα αυτές τις δημερίες δομές να τις μετασχηματίσουμε σε κάτι το οποίο θα έχει μια ευρωπαϊκή διάσταση και θα εξαρτάται λιγότερο από άμεσες διμερείς, έστω και πολυμερείς συνεργασίες και συμφέροντα των κρατών μελών. Δηλαδή, εντάξει, να διαθέσουμε τα χρήματα, αλλά από εκεί και πέρα πόσο ρεαλιστικό είναι ότι θα δημιουργηθεί αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση. Γιατί στην πολιτική συζήτηση Όλοι θέλουν να κάνουν την Ευρώπη, αλλά ακόμα και ο πρόεδρος Μακρόν, ο οποίος έδειξε πολύ μεγάλη φιλοδοξία, με την καλή έννοια, ε, σε λεπτομέρειες αν το δείτε, πάλι διμερή συνεργασία θέλει ή πολυμερή μεταξύ κρατών. Πόσο ρεαλιστικό λοιπόν είναι να έχουμε αυτή την ευρωπαϊκή προσέγγιση. Και μια τελευταία ερώτηση. Σε σχέση με αυτά που είπε ο κύριος Τόμα για την αριστεία καθηγητής, στην έρευνα για τα θέματα ασφαλείας, αλλά και σε πολλά άλλα θέματα, η αριστεία είναι κάτι ε, το οποίο είναι σχετικά ε, εύκολο να ελεγχθεί, να αποδειχθεί. Αλλά όταν μιλάμε για κοινέ προμήθειες, ένα νέο σύστημα ε, ευρωπαϊκό, η αριστεία είναι κάτι το σχετικό και πώς μεταφράζεται εκεί αφού μέχρι τώρα ε, οι κυβερνήσεις είναι αυτές που κάνουν κρατικές προμήθειες κάθε φορά και ε, η προτίμηση δεν ήταν κάθε φορά με βάση την αριστεία ποιος έχει το καλύτερο προϊόν αλλά υπάρχουν και άλλες σκοπιμότητες πολιτικές, διμερείς, εθνικές τώρα κάνουμε κανένα ποιοτικό άλμα ή υπήρχε αυτή η αριστεία από πριν και πώς ορίζεται Και ήταν ένας από τους βασικούς στόχους, μάλλον αρχές, ε, των ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Αλλά δεν ταυτίζεται απόλυτα με την εκάστοτε εθνική αμυντική έρευνα που είχε άλλο προσανατολισμό τα εθνικά συμφέροντα, αλλά όχι πάντα την αριστεία ως γνώμονα. Πριν δώσω το λόγο στον επόμενο Έχουμε δύο συντονιστές στην αίθουσα. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Κύριε Έλλερ, από όσο γνωρίζω, είμαι η μόνη πολιτικός εδώ με εμπειρογνώμονες για την έρευνα στην άμυνα που μιλούμε για την σημερινή κατάσταση της ανάπτυξης της αμυντικής βιομηχανίας, αλλά και τις εξελίξεις στην έρευνα για την άμυνα. Γνωρίζουμε ότι είμαστε πρωτοπόροι. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε τις παρουσιάσεις και για οποιονδήποτε πολιτικό είναι σαφές ότι είναι πολύ ενδιαφέρον το επίπεδο ανάπτυξης θα έλεγα μάλιστα και το επίπεδο συντονισμού μεταξύ των ε, ευρωπαϊκών ε, θεσμών και σε σχέση με το εθνικό επίπεδο, τη κατάσταση επικρατεί δηλαδή στο εθνικό επίπεδο. Τώρα για να σχολιάσω για τη δικιά σας πολιτική ερώτηση, γιατί καταλαβαίνω ότι οι πολιτικές ε, ερωτήσεις απευθύνονται εδώ στο βήμα, άρα στους πολιτικούς και επειδή είμαι μόνη πολιτικός εδώ στο βήμα αυτό, γι' αυτό απαντάω. Λοιπόν, την ευθύνη την έχει το Συμβούλιο. Και σας παρακαλώ, μην χαλάτε τον χαρακτήρα πραγματομοσύνης που έχει η συνάντηση αυτή. Είναι πολύ σημαντικό για μας να εκτιμήσουμε ποια είναι η κατάσταση στην αμυντική έρευνα και γι' αυτό αυτό σας παρακαλώ να αντιμετωπίσετε με τον ίδιο τρόπο όλους. Κύριε Γκάλερ τώρα. Ο κύριος Ελρά απαντάει. Κοιτάξτε, δεν θα αποφασίσετε εσείς τι θα ρωτήσω και τι όχι. Μπορεί για σας να είναι στο δικό σας το μυαλό ότι κάνω ερμηνεία, πολιτική κτλ. Αλλά δεν είναι έτσι. Εγώ απλώ ρωτώ. υπάρχει κάποιο εθνικό πρόγραμμα το οποίο να συνδέεται με αυτή την κοινή ιδέα για κοινή έρευνα. Αν δεν υπάρχει εθνικό, τότε είναι απλώς μια ερώτηση. Είναι θέμα εθνικής στρατηγικής ή όχι. Γιατί δεν έχει νόημα να φτιάχνουμε έρευνα αν δεν αποτελεί μέρος μιας κοινή στρατηγικής. Αυτό λέω απλά. Και είναι ερώτηση και για τους άλλους. Υπάρχουν εθνικές στρατηγικές οι οποίες να συνδέονται με αυτό που κάνουμε στον ε, τομέα της άμυνας και δεν έχει καμία σχέση με το Συμβούλιο. Είναι μια πρακτική ερώτηση. Αν εσείς αναφέρεστε στη χώρα σας, εντάξει, πολύ καλά κάνετε αλλά ας δούμε τις στατιστικές. Αν κοιτάξουμε τι συμβαίνει στις 28 χώρες ε, μέλη και πούμε ότι 12 έχουν εθνική στρατηγική που θα μπορούσε να ανταποκριθεί κάλλιστα για να αναπτυχθεί η ερευνητική τους δυνατότητα και οι υπόλοιπε δεν έχουν, για διαφορετικούς λόγους η καθεμία, είναι θεμετό το ερώτημα. Στους προσκεκλημένους μας που μας μιλάνε για τις ερευνητικέ φιλοδοξίες της άμυνας. Υπάρχει λοιπόν ρωτάω ένα πλαίσιο στην εθνική πολιτική. Δεν είναι το Συμβούλιο που θα κάνει οποιαδήποτε ερμηνεία. Είναι μια απλή ερώτηση και για τη Γερμανία και για την Πολωνία και για τις 28 χώρες. Αν πρέπει να ε, δαπανίσουμε στην αμετική έρευνα εφόσον δεν υπάρχει πλαίσιο κοινό πλαίσιο που έχει να κάνει με την ολοκλήρωση στην Ευρώπη. Είναι μια πρακτική ερώτηση και χερμηνίας. Για να ξέρουμε στην πράξη τι γίνεται με αυτές τις δραστηριότητες. Η Πρόεδρος. Εντάξει, υπονοήσατε κάτι, αλλά τέλος πάντων. Να εξηγήσω κι εγώ γιατί έχουμε εδώ αυτό το πάνελ. Δεν γνωρίζω κανένας από τις ομιλητές μας να είναι υπεύθυνο για εθνικές επιλογές και για εθνικά προγράμματα. Ίσως θα ήταν προτιμότερο την ερώτησή σας να την ε, υποβάλλετε στο απογευματινό μας πάνελ με θέμα το μέλλον της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Άμυνας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Γιατί εκεί θα μπορούσαμε να το ρωτήσουμε και να καλέσουμε και πάλι τον κύριο Τόμεκ, άμα θέλετε, ή την Επίτροπο Βγόσκα και άλλους από την Επιτροπή, την ε, Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και να ρωτήσουμε αυτούς ποιο είναι το επίπεδο συντονισμού. Αυτοί πρέπει να απαντήσουν σε αυτό και όχι οι πυρογνώμονες. Εν πάση περιπτώσει, έχετε δικαιώμα να ρωτάτε ό,τι θέλετε, αλλά νομίζω ότι οδηγεί σε παρεξηγήσεις. Κύριε Γκάλερ, εσείς τώρα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι και τους τρεις σας που ελπίζετε ότι μπορείτε να υποφεληθείτε από ευρωπαϊκά κονδύλια και μετά η ευρωπαϊκή πλευρά εκείνη θέλει να ενισχύσει τη συνεργασία όταν δίνει κονδύλια για την έρευνα στην άμυνα. Όπως έχουν τα πράγματα σήμερα, βλέπετε εσείς προβλήματα για χρηματοδότηση όταν συνεργάζεστε μεταξύ σας πιστεύετε ότι υπάρχει ανάγκη να βελτιωθεί ο τρόπος που δρά η Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να σας διευκολύνει, να έχετε χρηματοδότηση για συμφωνημένη συνεργασία μεταξύ σας. Ή έτσι όπως έχουν τα πράγματα σήμερα και σε άλλους τομείς έρευνας, πιστεύετε ότι για την αμυντική έρευνα ειδικότερα υπάρχουν προβλήματα για να φτάσουν στα χέρια σας ε, τα κονδύλια, η χρηματοδότηση. Πρόεδρος, ο κύριος, κυρία Λόζινγκ είναι η επόμενη συντονίστρια, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ γερμανικά μιλώ. Μάλιστα. Όλα αυτά που μας παρουσιάσατε και δεν θέλω να μπω καθόλου τώρα στις τεχνικές λεπτομέρειες. Θα ήθελα να τα σχολιάσω υπό την πολιτική έννοια, σε ένα πολιτικό πλαίσιο να το συζητήσουμε. Είναι πάρα πολύ ευρύς ο τομέας αυτός, πάρα πολύ διασυνδεδεμένος, με πάρα πολλές διαφορετικές διαστάσεις. Χρηματοδότηση, έρευνα, παραγωγή, πώληση, στρατηγική, σχεδιασμός ο κύριος Έλερ μίλησε και για κοινέ προμήθειες αμυντικού υλικού. Και τώρα εμείς είμαστε ε, σε ένα χώρο που εξετάζει και προσωπεί την κοινοβουλευτική διάσταση. Και όπως συμβαίνει σε όλα τα κοινοβούλια και σε όλες τις πολιτικές ε, ομάδες και σχηματισμούς, υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευση, υπάρχει και η μειοψηφούσα άποψη. Και τι γίνεται τώρα για τη χρηματοδότηση της αμυντικής ε, έρευνας. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και υπάρχουν και επικριτικά βλέμματα. Κύριε Τόμα, εσείς μιλήσατε για το ρόλο της ομάδας προσωπικότητων. Και στο τέλος είπατε ότι εδώ μπορεί να συνεργαστεί όποιος θέλει και διαθέτει την ε, εν λόγω πραγματογνωμοσύνη και εμπειρία. Κοιτάω τη σύνθεση της ομάδας προσωπικότητων και τι διαπιστώνω. Έχει 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως για την άμυνα προτείνει ένα ταμείο, ας πούμε, που υιοθετήθηκε η πρόταση αυτή σχεδόν ατόφια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κάτι μου λείπει από τη σύνθεση της ομάδας προσωπικότητων. Θα ήθελα ένα ευρύτερο φάσμα. Και σας ερωτώ, έτσι ευθέως κύριε Τόμα, και τη δική σας οργάνωση που είπατε ότι εκπροσωπείστε εκεί στην ομάδα προσωπικότητων ε, στο πρόσωπο του του Διευθύνοντα Συμβούλου, δεν ξέρω πώς τον λένε. Ε, δεν το θεωρείτε προβληματικό αυτό? Ότι δεν υπάρχει καμία φωνή επικριτική εκεί, κανένα πρόσωπο στην ομάδα προσωπικότητων που να συνιστά μια αντιπολίτευση, μια διαφωνία, μια άλλη φωνή διαφορετική οι διάφοροι εκπρόσωποι και τα διάφορα μέλη σε αυτή την ομάδα προσωπικότητων εποφελούνται, έχουν οικονομικό όφελος άμεσο από αυτά που προτείνουν, έχουν οικονομικό συμφέρον. Μήπως το μέλλον χρειάζεται να είναι ευρύτερη η σύνθεση ενός τέτοιου οργάνου για να έχουμε και εκπροσώπους άλλων ε, ρευμάτων, ε, οργανισμών και μια φωνή αποκλίνουσα, εν πάση περιπτώσει. Ευχαριστώ. Thank you. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο, ο πρόεδρος, ο επόμενος. Επιτρέψατε μου να αναφερθώ σε κάτι που είπε ένας συνάδελφος. Μήπως παραβλέπετε το ότι σήμερα η κατάσταση έχει αλλάξει. Κατά τη γνώμη μου, η σημερινή κατάσταση χαρακτηρίζεται από τρεις μεταβλητές, τρία στοιχεία. 22 κρατημένα δεν κάνω λάθος, έχουν υπογράψει αυτή τη συμφωνία για την ΠΕΣΚΟ, την ε, μόνιμη διαρκή συνεργασία. Και η Πολωνία μεταξύ αυτών των χώρων είναι οι χώρες που ίδρυσαν, που συγκρότησαν αυτή την συνεργασία, την ΠΕΣΚΟ. Και από ό,τι φαίνεται, για πρώτη φορά μας δίνεται η ευκαιρία να υπάρχει κάλυψη από τον προϋπολογισμό. Για πρώτη φορά λοιπόν στην επόμενη χρήση θα υπάρχουν κονδύλια για την άμυνα και την ασφάλεια. Και κάτι άλλο τώρα, το οποίο επίσης δεν έχει προσεχθεί αρκετά. Για μένα πάντως είναι θέμα που με απασχολεί εδώ και χρόνια. Νομίζω ότι στην Ευρώπη δεν έχουμε συνειδητοποιήσει τόσο πολύ την διαφορά τεχνολογικής πρόοδου μεταξύ ημών και των ΙΠΑ. Ε, μιλάμε ότι είμαστε πίσω πέντε χρόνια γενικώ και όσον αφορά τα υλικά ίσως μια δεκαετία πίσω σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Η πρόοδος επίσης της Ρωσίας είναι εντυπωσιακή γιατί είχαν κολλήσει για ένα μεγάλο διάστημα οι Ρώσοι. Οπότε θα πρέπει να αφιερώσουμε περισσότερους πόρους για άμυνα και ασφάλεια εδώ στην Ευρώπη. Και επίσης να προσέξουμε το θέμα των νέων τεχνολογιών, την έρευνα και την εφαρμογή. Δεν αρκούν αυτά που αφιερώνουμε προς το παρόν. Επίσης θα πρέπει να δούμε εδώ στην Ευρώπη ποια είναι τα προγράμματα τα οποία μπορεί να χρηματοδοτηθούν από τον κοινωνικό προϋπολογισμό. Μιλούμε για δισεκατομμύρια ευρώ στο οποίο θα φτάσει το κόστος ε, σε λίγα χρόνια. Άρα, να δούμε ποιες είναι οι έρευνες που θα είναι επιλέξιμες σε κάθε κράτος. Και επίσης τι μπορούμε να κάνουμε από κοινό. Δεν γίνεται ο καθένας μόνος του να αναλάβει αυτόν τον ε, ρόλο. Άρα και σε πολιτικό και σε στρατικό επίπεδο πρέπει να ληφθούν κάποιες αποφάσεις. Και να δούμε τι θα πρικοδοτήσουμε. Ένα θέμα αυτό. Το δεύτερο. Εδώ έχουμε τρεις σπουδαίους εμπειρογνώμονες. Είναι εντυπωσιακέ οι γνώσεις τους. Και τους ε, ερωτώ Βέβαια και θα έχετε αναλύσει τι γίνεται στο Ισραήλ, στη ΣΥΠΑ, στη Ρωσία. Πεςτε μας ποιες είναι οι διαφορές ε, μεταξύ ημών και εκείνων. Ο κ. Γκάλερ θέλει το λόγο. Γερμανικά. Πάρα πολύ σύντομα για να διευκρινίσω αγαπητή συνάδελφε Λόζινγκ. Η χρονική σειρά με τα 500 εκατομμύρια πώς έχει στην ομάδα προσωπικότητων, ακούστηκε αυτό το νούμερο, μετά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά πλειοψηφία το υπερψήφισε, τα 500 εκατομμύρια είναι η λιμένη απόφαση του Κοινοβουλίου και μετά ήρθε η Ευρωπαϊκή Επίτροπη και το πρότεινε. Παρακαλώ να μην διαδίδουμε εδώ πέρα παραμύθια ότι υπάρχει καμιά σκοτεινή δύναμη ομάδα προσωπικότητων που ασκεί πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και φυτεύει εκεί τα συμφέροντά της. Δεν το υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από εκεί πρώτα αποφασίστηκε από το Κοινοβούλιο για να ξέρουμε ποια είναι η χρονική αλληλουχία όλων αυτών. Ευχαριστώ. Κύριος Κρασνοντέμσκι. Ε, ε, Εγώ με τη σειρά μου να σας ευχαριστήσω. Ήταν πολύ ενδιαφέροντα τα όσα ακούσαμε από εσά. Ήταν πολύτιμη αυτή η ενημέρωση. Ο κύριος Τωμά Ναι, αυτά που είπε κάπως με κάνει αισθάνομαι απεσιόδοξος. Μας δείξατε δύο χάρτες. Πρώτα-πρώτα ήταν ένας ε, χάρτης για το Ίδρυμά σας στην ε, Γερμανία. Και εκεί απεικονιζόταν η νοτιοανατολική Γερμανία. Όχι, συγγνώμη, συγγνώμη, βόρεια Ανατολική Γερμανία διορθώνει. Ήταν λοιπόν μια λευκή ζώνη εκεί στον χάρτη της Γερμανίας. Στη συνέχεια μετρήσατε ένα χάρτη της Ευρώπης. Εκεί απεικονίζατε τα ιδρύματα που ασχολούνται με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία και είδαμε ότι υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση από τέτοια ιδρύματα ε, σε συγκεκριμένες περιοχές, ας πούμε στον πυρήνα της Ευρώπης. Εντάξει, είναι τόσο μυστήριο, εξηγείται γιατί έχουμε τόσο υψηλή ποιότητα έρευνα στις γεννημένες περιοχές και ξέρουμε ότι και με το ορίζον 2020 υπάρχουν θέματα, υπάρχουν προβλήματα, κάποια κρατημέλη τα οποία εισφέρουν, αλλά όχι άλλα, υπάρχει δηλαδή έλλειψη ισορροπίας, οπότε σας παραπέμπω και σε αυτά που έξω από τον κύριο Έλερ όσον αφορά τους στόχους των εν λόγω προγραμμάτων είναι και πολιτική η στόχη των προγραμμάτων. Α, το είδε και το πεσήμενο και ο κύριος ε, Γιούγκερ που για την αύξηση της ε, στρατιωτικής συνεργασίας στον τομέα της άμυνας που θα πρέπει να μας βοηθά στον ε, τομέα, στο μέτωπο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Οπότε ακριβώς βλέποντας την άνισορροπία στο ιστορικό της Γερμανίας βλέπουμε ότι και στο ιστορικό της Γερμανίας υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά ε, την ε, ολοκλήρωση, όσον αφορά την εξισορρόπηση ε, ανατολικής με δυτικής Γερμανίας. Πάντα μιλάμε για τον τομέα τώρα της επιστημονικής έρευνας. Οπότε, αν σε 10 χρόνια έχουμε την ίδια απεικόνηση, την ίδια κατάσταση στο χάρτη, τότε αυτό σημαίνει πρόβλημα. Σημαίνει ότι είναι δύσκολο να πετύχουμε τους τεθέντες στόχους. Δεν θα έχουμε βελτιώσει τις ευρωπαϊκές δυνατότητες θα πρέπει να υπάρχει πιο εξορροπημένη ανάπτυξη στην Ένωση. Θα πρέπει να υπάρξει περισσότερη ελεγγύη. Γιατί η ισορροπία και στην πρόοδο της τεχνολογίας πάει να πει και αλληλεγγύη. Και γι' αυτό τα κρατη από Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη έχουν πολλές επιφυλάξεις για όλα αυτά τα προγράμματα, για όλα αυτά τα πλάνα ε, είναι, είναι δύσπιστα τα κράτη αυτά, τα μέλη αυτά, επειδή δεν υπάρχει αυτή η ισορροπία. Εσεί πέστε μα λοιπόν, μια που είστε επιστήμονε που εργάζεστε σε αυτό το τομέα, τι θα μπορούσε να γίνει για να γεφυρωθούν αυτά τα κενά, αυτή η απόσταση. Ο κύριο Λίτ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά κι εγώ. Κύριε Πρόεδρε, καταλαβαίνετε γερμανικά. alles klar. Also, I Μπορώ να μιλήσω για αγγλικά, άμα θέλετε. Θα ήθελα να πω κάτι γενικό. Ένα συνάδελφός μου ρώτησε κάτι το πάνελ. Δεν είναι συζήτηση μεταξύ των εμπειρογνωμόνων στο πόντιουμ. Είναι μια συζήτηση που κάνουμε στην Επιτροπή μας επί της ουσίας. Και όταν κάνουμε πολιτικές ερωτήσεις θα πρέπει να διατηρήσουμε ανοιχτό το πνεύμα μας εδώ, να μπορούμε να κάνουμε και πολιτικές ερωτήσεις που έχουν σχέση με πολιτικά ζητήματα ευρωπαϊκά και να μην επικρίνουμε συναδέλφους που κάνουν ερωτήσεις εμπειρογνώμονες. Δεν συζητάμε με το Συμβούλιο εδώ. Μια ειλικρινή απάντηση θέλω να δώσω στο συνάδελφο που ρώτησε για το Ινστιτούτο Φρόνχοφερ. Εγώ είμαι από την Ανατολική Γερμανία και εκεί εργάζεται για τις νέες τεχνολογίες και τις νέες επιστήμες, ε, την τεχνολογική επανάσταση 4.0. Έχουμε και στην Ανατολική Γερμανία καλά Ινστιτούτα τεχνολογικά. Μπορεί να είναι λιγότερα, αλλά είναι ευρύτερη η ε, σύνδεση και η δικτύωση. Έχουμε δύο Ινστιτούτα, Fraunhofer, ε, πολύ μεγάλα. Μην ανησυχείτε. Επί της ουσίας τώρα εργαζόμαστε σε ένα τομέα που για μένα ως Γερμανός, ως είναι εύκολο να το ε, καταλάβω σε μακροχρόνια προοπτική και σας ευχαριστώ που διοργανώσατε αυτή την ακρόαση γιατί θέλουμε οι Γερμανοί σοσιαλδημοκράτες να δημιουργήσουμε στρατιωτικές δυνατότητες και ικανότητες και ε, ε, για έναν ευρωπαϊκό στρατό αλλά και για pooling and sharing, δηλαδή συνένωση και κοινή ε, χρήση των ικανοτήτων των στρατιωτικών που έχουμε. Έχουμε τώρα μια ευκαιρία για την άμυνα και τη χρηματοδότηση που μπορεί να είναι χαμηλότερη από εκείνη που θα προτιμούσαμε. Το θέμα είναι πώς θα προχωρήσουμε τώρα εμείς, αλλά και τι θα κάνουν τα κράτη-μέλη για να μας δώσουν ένα πλαίσιο και να έχουμε κάτι να πούμε, γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είναι και πάγια θέση του κόμματός μου, πρέπει να έχει μεγαλύτερο λόγο για θέματα της υποεπιτροπής μας και αυτό αφορά και ε, την παραγωγή όπλων και την εξαγωγή όπλων που είναι όλα αυτά αλληλένδετα. Λοιπόν, έρευνα και εξαγωγές αμυντικού υλικού. Ποια είναι η εμπειρία της γαλλογερμανικής συνεργασίας για τα προϊόντα που έχουμε αναπτύξει και πώς τα εξάγουμε και πώς πηγαίνουν οι εξαγωγές μας. Είναι ενδιαφέρον αυτό. Ένα συνάδελφός μου παρακολουθεί τα όσα συζητούν οι Μακχόν και Μέρκελ ε, για την παραγωγή αλλά και την εξαγωγή, επαναλαμβάνω, εξαγωγικές ε, δομές. Έχω και μια ερώτηση για την Πολωνία, από τον εκπρόσωπο από την Πολωνία. Ποιε είναι οι ευρωπαϊκέ χώρε με τι οποίες συνεργάζεστε και συζητάτε για εξαγωγές ε, των προϊόντων που αναπτύσσετε. Προφανώς στην άμυνα κυρίω. Και για τον κύριο Τόμα θέλω να ρωτήσω. Υπάρχουν θεσμοί, ερευνητές, πανεπιστήμια, Ινστιτούτα στην Ανατολική Ευρώπη που συνεργάζονται στον τομέα σας. Ευχαριστώ πολύ. Um, Ευχαριστούμε. Για να απαντήσω σε ό,τι με αφορά τουλάχιστον. Η δικιά μου παρέμβαση έγινε επειδή ρητά αναφέρθηκε η χώρα μου και δεύτερον σε ένα πολιτικό πλαίσιο. δεν είχε να κάνει με το περιεχόμενο του πάνελ. Είσαστε μάλλον νέος στην Επιτροπή αυτή, καλώς ήρθατε, αλλά τρία χρόνια εδώ προσπαθούμε να έχουμε υψηλού επίπεδου πραγματογνωμοσύνη και αυτό ακριβώς κάνει και το σημερινό μας πάνελ. Αυτή την ιδέα καλύπτει. Και συζητούμε σε επίπεδο πραγματογνωμοσύνης. Όταν έχουμε πολιτικά ζητήματα, τότε καλούμε αξιωματούχους των ευρωπαϊκών ε, οργάνων υψηλού επίπεδου, έτσι, και τότε συζητάμε πολιτικά θέματα. Τώρα, ο κύριος Πουστινάρο έχει το λόγο, νομίζω. Κύριε Άλλερ, θέλετε διαδικαστικό. Ναι, μια ερώτηση διαδικαστική. Νομίζω μέχρι την επόμενη φορά θα πρέπει να διευκρινίσουμε και για την Πρόεδρο ότι λέει ο κανονισμός. Πού λέει ο κανονισμός ότι μπορεί η Πρόεδρος να ερμηνεύει, ποιες ερωτήσεις είναι πολιτικές, ποιες κάτι άλλο και σε ποιο βαθμό μπορούν ή πρέπει να απαντήσουν οι προσκεκλημένοι. Στο βαθμό που όλοι οι παρόντες είναι ενήλικες μπορεί κάποιος επισκέπτης να πει ότι αυτό το θεωρώ πολιτική ερώτηση. Εγώ είμαι υπερογνώμων ε, και δεν είμαι σε θέση, δεν είμαι πρόθυμο να το απαντήσω. Στον κανονισμό του Κοινοβουλίου εγώ δεν βλέπω πουθενά που να λέει ότι μία πρόεδρος θα μπορούσε να τολμήσει να ερμηνεύσει τι ε, μπορούν ή τι επιτρέπεται να απαντήσουν προσκεκλημένοι εμπειρογνώμονες. Οι άνθρωποι είναι ενήλικες, εκπροσωπούν ε, θεσμούς και βεβαίως έχουν μια αυτοπεποίθηση, έχουν γνώση, έχουν εμπειρία και είναι σε θέση να αποφασίσουν τι θέλουν, τι μπορούν και τι επιτρέπεται να απαντήσουν. Μπορείτε να μου δείξετε στον κανονισμό ποιο είναι το δικαίωμα της Προέδρου να κάνει διάκριση, ποιες ερωτήσεις είναι πολιτικές, μη πολιτικές, αμφισβητήσιμες ή όχι, να μου το πείτε. Εάν μέχρι την επόμενη φορά δεν μου το έχετε διευκρινίσει ότι προβλέπετε από τον κανονισμό, θα προτείνω, θα παρακαλέσω την Πρόεδρο να μην κάνει τέτοια πράγματα. Αλλιώς να κάνουμε καμιά ψηφοφορία εδώ, αν δεν μπορεί η Πρόεδρος να τηρήσει τον κανονισμό, μήπως είναι ακόμα ενδεδειγμένη Πρόεδρος της Υποεπιτροπής μας. Πρόεδρος. Νομίζω ότι σίγουρα θα έχουμε σύντομα διευρυγμένο Προεδρείο και μπορείτε να θέσετε αυτό το ζήτημα στο διευρυμένο Προεδρείο. Η παρέμβασή μου ήταν ακριβώς επειδή αναφερθήκατε στη χώρα μου και χρησιμοποίησατε τον όρο πολιτικό, political. Γι' αυτό και παρενέβη. Ο κύριος Μποστινάρου τώρα. Ευχαριστώ. Επιτέλους, κύριε Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις έχω. έχοντα ακούσει τους τρεις εξέχοντες εμπειρογνώμονες. Πρώτον, πώς διασφαλίζουμε και τι ρόλο πρέπει να παίζουν οι χώρες μέλη που εμπλέκονται σε κοινά σχέδια αμυντικής έρευνας για να αποφευχθούν ανισορροπίες. Γιατί όπως είδαμε και στο Γιούκαρς, ενώ όλοι συνεισφέρουμε ή ενώ υπάρχει μεγάλη δέσμευση. Η Ρουμανία, για παράδειγμα, ήδη συμμετέχει στην ΠΕΣΚΟ. Η Ρουμανία ε, θέλει να ασχοληθεί, αλλά στο μέλλον να μην γίνει αυτό που έγινε και με το σχέδιο Juncker και εδώ στην έρευνα και την ε, τεχνολογία στην άμυνα, Οπότε ο σχεδιασμός προβλέπει εγγυήσει για δίκαια συμμετοχή σε τέτοια κοινά προγράμματα, λαμβάνοντας υπόψη και τον ρόλο τους στη συντήρηση. Γιατί φυσικά καμία χώρα δεν μπορεί από μόνη της να γίνει ένας μεγάλος αμυντικός παραγωγός. Δεύτερον, θα ήταν καλύτερα να αρχίσουμε με μικρότερα προγράμματα, μικρότερες κλίμακας. Τα cyber, hybrid, drones, όπου συνεργαζόμενοι μπορούμε να βελτιώσουμε την αδύναμη ικανότητα που έχουμε και έτσι να κερδιθεί εμπιστοσύνη και να προωθήσουμε στη συνέχεια την έρευνά μας και σε πιο σημαντικά προγράμματα. Μήπως γιατί δεν βλέπω πώς θα αποφύγουμε μεγάλη αμυντική παραγωγή, ε, πώς θα το αποφύγουμε να γίνουν ακόμα μεγαλύτερη και τελικά η ευρωπαϊκή ε, άμυνα να μείνει στο περιθώριο. Αυτό πρέπει να φροντίσουμε με τη συνεργασία μας. Επίσης αναφερθήκατε στη στρατηγική αυτονομία. Ωραίο είναι, αλλά ακριβώς εδώ σε αυτή την αίθουσα έχουμε ακούσει έναν εξέχοντα Γάλλο διπλωμάτη, δεν θα πω ποιο ήταν, ο οποίο είπε ότι η στρατηγική αυτονομία δεν είναι ρεαλιστική. Και με την λίγη γνώση που εγώ έχω, προκειμένου να έχουμε στρατηγική αυτονομία, πρέπει να έχουμε μια πραγματικά κοινή αμυντική στρατηγική. Στη σημερινή πραγματικότητα υπάρχουν προκλήσεις ασφάλειας και άμυνας διαφορετικές στην Ανατολή, στον Νότο κλπ. Οπότε η άμυνα και η ασφάλεια δεν είναι μόνο αποστολές πέσκο σε διάφορα μέρη της Αφρικής ή της Μέσης Ανατολής, είναι κάτι παραπάνω. Είναι πραγματικά η ικανότητα να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Γιατί τι σημαίνει η κοινή ε, πολιτική. Σημαίνει να είμαστε έτοιμοι να φέρουμε σε πέρα σε ένα πόλεμο, όχι μόνο να μιλάμε για αυτόν. Και πολύ θα το ήθελα. Μπορούμε να πάμε προς αυτή την κατεύθυνση προκειμένου να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε άμυνα, ασφάλεια και κοινή άμυνα και ασφάλεια, στρατηγική δηλαδή κοινή άμυνα και ασφάλειας προκειμένου να έχουμε μια κοινή στρατηγική και στρατηγική αυτονομία, με μία όμως παρατήρηση. Η στρατηγική μας αυτονομία και όλο το στρατηγικό κεφάλαιο στο οποίο θα καταλήξουμε, ποτέ δεν θα πρέπει να είναι σε ανταγωνισμό με το ΝΑΤΟ. Δεν θα πρέπει ούτε να θέλει να ε, αποσχεστεί από το ΝΑΤΟ, αντίθετα να φροντίζει πάντα να υπάρχει συμβατότητα και διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Κύριε Μποστινάρο, τέλειωσαν οι ερωτήσεις και απαντήσεις και τώρα να απαντήσουν ε, οι εμπειρογνώμονές μας, οι προσκεκλημένοι μας στις ερωτήσεις και στα σχόλια. Και αρχίζουμε με τον κύριο Ντιλεβαλμένη. Ευχαριστώ. Δύσκολο να απαντήσω τόσες πολλές ερωτήσεις. Ε, θα προσπαθήσω, αν και είναι πολλές. Θέλω να έρθω στις τελευταίες ερωτήσεις που κάνατε. Ή μάλλον πρώτα απ' όλα να πω ότι εγώ εδώ εκπροσωπώ το Γαλλογερμανικό Ινστιτούτο Ερευνών, γαλλική άμυνα, όχι τόσο γερμανική, αλλά για να έρθω στην τελευταία σας ερώτηση. Σήμερα δεν μιλάμε για την προμήθεια ικανοτήτων για την προσφορά ικανοτήτων. Μιλάμε για την έρευνα και την τεχνολογία. Την προσφορά αυτών των δύο. Όταν λέτε πώς θα αποφύγουμε τις ανισορροπίες, δεν μπορούμε να γνωρίσουμε το γεγονός ότι διάφορες χώρες μέλη επενδύουν εδώ και χρόνια στην έρευνα και την τεχνολογία και συνεχίζουν και το κάνουν πολύ περισσότερο από ό,τι άλλες. Αυτό είναι ένα γεγονός. Τώρα, Σε μερικές από αυτές τις χώρες μέλη υπάρχουν κέντρα αριστείας, τα οποία θα έπρεπε να χρησιμοποιούνται ώστε συλλογικά να προθούμε την αμυντική μας έρευνα και τεχνολογία. Στην παρουσίασή μου είπα με ποιο τρόπο το κάνουμε εμείς, πώς εργαζόμαστε δηλαδή. Γιατί κάποιος είπε μπορούμε να εξευρωπήσουμε το ε, Ινστιτούτο αυτό. Πριν από λίγα χρόνια προσπαθήσαμε να έχουμε τέτοιες συνεργασίες και δεν πέτυχε γιατί ετοιμάστηκε από πάνω προς τα κάτω. Αυτό που τώρα προσπαθούμε να κάνουμε είναι από κάτω προς τα πάνω να πετύχει αυτός ο εξωευρωπαϊσμός. Πώς θα γίνει. Είναι αυτό που εξήγησα και πριν. Ότι δηλαδή στο δικό μας τομέα αριστείας και πραγματογνωμοσύνης έχουμε χρηματοδότηση εδώ και χρόνια και πιστεύω ότι πάμε πολύ καλά. Είμαστε ένα κέντρο αριστείας. Όμως, εκτός από τους ανθρώπους που έχουμε, Χρειαζόμαστε και εμπειρογνώμονες από άλλες χώρες. Και για παράδειγμα έχουμε συγκεκριμένου χρόνου συμβάσεις και κάποιες από αυτές τις συμβάσεις είναι από τη δική σας χώρα. Οι άνθρωποι αυτοί λοιπόν που είναι πολύ καλοί επιστήμονες εποφελούνται έτσι από τη δικιά μας υποδομή, εποφελούνται από την διεθνή ατμόσφαιρα, το διεθνές κλίμα που επικρατεί στο Ινστιτούτο μας και στο τέλος της σύμβασής τους θα επιστρέψουν στη χώρα σας, στη χώρα τους και θα συνεχίσουν την έρευνα και την τεχνολογία στον τομέα της άμυνας. Και αυτό που ισχύει για την Ρουμανία, ισχύει και για την Πολωνία, για τη Λιθουανία, για όλες τις χώρες με τις οποίες έχουμε στρατηγικές συμφωνίες με επιστημονικά Ινστιτούτα και εδώ ο Πολωνός συνάδελφος το γνωρίζει. Πρέπει να ομολογήσω ότι μέχρι τώρα δεν ήξερα ότι υπήρχε το ΡΙΑΠ. Ομολογώ. Το ΠΙΑΠ, συγγνώμη. Το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Ερευνών Αρθωματισμού και Μετρήσεων. Να λοιπόν, πεδία συνεργασίας που μας περιμένουν και θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Για τα μη επανδρομένα δεν το κάνουμε μέχρι τώρα. Θα μπορούσαμε. Πώς θα αποφύγουμε ή θα μειώσουμε τις ανισορροπίες, ρωτάτε. Αυτό δεν είναι κάτι το οποίο έρχεται και επιβάλλεται από πάνω. Θα έπρεπε Αυτό τι σημαίνει, σημαίνει ότι τελικά όλοι θα προχωρήσουμε στην αμυντική έρευνα και τεχνολογία. Για την ερώτησή σας για τις εξαγωγές. Έχουμε κάτι καλό στο Ινστιτούτο μας που είναι γαλλογερμανικό. Ξέρετε ότι οι εξαγωγές είναι εθνικό θέμα για αμυντικά προϊόντα, ακόμα και έρευνα και τεχνολογίες. Οπότε γινόμαστε Γάλλοι όταν πρέπει και Γερμανοί όταν πρέπει, ανάλογα. Και αυτό είναι κάτι που λειτουργεί και βοηθάει πολύ. Βάζουμε το καπέλο του Γερμανού το καπέλο του Γάλλου, ανάλογα. Τώρα για τις διάφορες παρατηρήσεις και ερωτήσεις που κάνατε. Και ο καθηγητής Τωμά αναφέρθηκε. Μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε με όλα όσα είπε ο καθηγητής Τομά. Υπάρχει συμφωνία από αυτόν αυτό που εγώ προσπάθησα να κάνω στη δική μου παρουσίαση και χτίζοντας πάνω στην ήδη υπάρχουσα συνένεση, τι μπορούμε να κάνουμε δηλαδή στα χαμηλά επίπεδα, από κάτω προς τα πάνω, για να βελτιώσουμε την έρευνα και την ε, τεχνολογία άμυνα στην Ευρώπη. Ευχαριστούμε ο καθηγητής ε, Σίνκαρτ. Κυρίες και κύριοι, Θα προσπαθήσω να σας απαντήσω. Έχουμε πολλές ερωτήσεις και δεν ξέρω αν θα μπορέσω όλους να σας καλύψω. Οπότε πρώτα πρώτα κάτι γενικότερο. Να τοποθετηθώ όσον αφορά αυτή την δύσκολη ερώτηση. Νομίζω ότι είμαστε σε δύσκολη θέση με οι επιστήμονες τώρα που βρισκόμαστε και έχουμε γύρω-γύρω τόσους πολιτικούς. Στην αρχή ε, έλεγα να πω ότι επιστήμονας είμαι, τι, τι να σας ε, απαντήσω. Όμως κάτι, που, κάτι που είναι σχεδόν προσωπική απόψη. Όταν προσχώρησε στην Ένωση η Πολωνία και όταν επίσης προσχωρήσαμε στην υπηρεσία διαστήματος, τότε θεωρήσαμε ότι μας ξανήγεται μία πόρτα, μία πύλη, ε, είναι κάτι που το περιμέναμε και οι επισκέπτες, ε, οι εταίροι μας επίσης θεώρησαν ότι υπάρχει ενθουσιασμός ε, άκρατος και αφορούσε ακριβώς αυτή την ευκαιρία μας και γι' αυτό σας διαβεβαιώνω ότι μας ενθουσιάζει αυτή η συνεργασία με τους Ευρωπαίους συναδέλφους. Και στην περίπτωση, επομένως, της ε, άμυνας και της ε, ασφάλειας. ότι προσφέρουμε τις γνώσεις μας ούτως ώστε να βελτιωθεί η διεθνή συνεργασία σε αυτούς τους τομείς και νομίζω ότι τα πάμε όλο ένα και καλύτερα. Ιδίως για την ασφάλεια. Ίσως ε, η άμυνα είναι περισσότερη υπόθεση και των πολιτικών, αλλά η ασφάλεια είναι κάτι που απασχολεί τους πάντες. Το έγκλημα, η τρομοκρατία, όλες οι, οι χώρες έχουν ε, προβλήματα. Και κάθε φορά που χρησιμοποιήθηκε ένα δικό μας ρομπότ σε κάποια πετυχημένη αποστολή, ακόμα και αν καταστράφει η επιτυχία της αποστολής, εμείς αισθανόμαστε ευτυχείς που η δουλειά μας έπιασε τόπο και ωφέλησε κάποιους. Δεν μπορώ να σας απαντήσω στο πολιτικό επίπεδο. Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας. Ελπίζουμε ότι τα πάμε καλά και ότι εξασφαλίζουμε καλύτερη άμυνα και καλύτερη ασφάλεια. Πάμε τώρα παρακάτω για τις άλλες ερωτήσεις. Ίσως η Ευρώπη έκανε μια σωστή κίνηση. Όταν αποφάσισε ότι κάποια θέματα θα τα αναλάβουν οι εθνικές υπηρεσίες πληροφοριών και να κάτσουν να δούνε ποιο μπορεί να εξειδικευτεί σε τι ανάλογα με τι ικανότητέ του. Αυτό ήταν μια τέτοια προσέγγιση από κάτω προ τα πάνω για να μην ανακατεύονται όλοι με όλα. Ε, τέτοια ανάλυση θα πρέπει να υπάρχει. Και έτσι θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε και σε εθνικέ αλλά και σε ευρωπαϊκέ στρατηγικές τώρα το τι μπορούμε να κάνουμε για καλύτερη πρικοδότηση των προγραμμάτων. Ο ανταγωνισμός χρειάζεται. Και αν έχουμε διάφορα ε, δίκτυα ε, τα οποία προσπαθούν να αποσπάσουν γνωμοδότηση για τα δικά τους προγράμματα, τότε θα έχουμε κάποιο ανταγωνισμό και τελικά θα ωφεληθεί αυτός που τα καταφέρνει καλύτερα. Άλλη ερώτηση αφορούσε τις διαφορές μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών και επίσης Ισραήλ αλλά και Ρωσία. Σας τα είπα στην εισηγησή μου ότι για το δικό μου τομέα όσον αφορά δηλαδή αυτά τα μη επανδρομένα οχήματα εδάφους θεωρούμε ότι πρόσφατα έκανε εντυπωσιακά βήματα πρόοδου η Ρωσία για αυτά τα οχήματα που χρησιμοποιήθηκαν στη μάχη. Το τόνισα. Επίσης, το Ισραήλ και η ΙΠΑ επίσης είναι πρωτοπόροι, προοδεύουν ταχαίως και αυτό για δύο λόγους. Πρώτα-πρώτα διαθέτουν πολλά χρήματα για αυτό το σκοπό. Και τα χρήματα αυτά τα διαθέτουν έτσι ώστε να πιάσουν τόπο. Έχουν αναλυθεί σωστά τα θέματα και αυτό αφορά και κάποιες άλλες ερωτήσεις για το κατά πόσο θα έχουμε μεγάλα προγράμματα ή μικρότερα. Να. Να σας πω από πλευράς κάποιου που φτιάχνει ρομπότ για αστυνομία, συνοριοφυλή κλπ. Έχουμε σχεδιάσει κάποια πολύ καλά ρομπότ από πλευράς μηχανικής είναι πάρα πολύ καλά. Τώρα από πλευράς του χρήστη θα μπορούσαν αυτά τα ρομπότ να καταστούν άχρηστα, να είναι άχρηστα και αυτό θέλω να σε εξηγήσω. Ότι εάν θέλουμε κάτι να φτιάξουμε θα πρέπει να ξέρουμε τι ζητάει, τι έχει ανάγκη ο χρήστης. Οπότε το ερώτημα που ανακύπτει είναι ποιος είναι ο χρήστης. Χρειάζεται μόνος να υπάρχει ένας πλήρης, σοβαρός διάλογος μεταξύ σχεδιαστών των προϊόντων μας και των χρηστών. Αλλιώς δεν βγαίνει τίποτα. Οπότε, να ξεκινήσουμε με κάποια μικρότερα προγράμματα. Οπότε με αυτό το προγράμμα να καλύπτουμε και την παραγωγή κάποιων προϊόντων αλλά και να ενθαρρύνουμε για τη συνεργασία με τους χρήστες. Άλλη ερώτηση ήταν το με ποιες χώρες συνεργάζεται το Ίδρυμά μας. Τι να σας πω, με όλες τις χώρες, με όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει καμία εξαίρεση. Να, με γίνει το πρόγραμμα Τάλος, για το οποίο σας μίλαγα, είχαμε εταίρους και από Τουρκία και από Ελλάδα. Ακριβώς σε μια φάση που υπήρχαν προστριβές μεταξύ αυτών των δύο χώρων. Όμως το πρόγραμμα είχε αίσια κατάληξη. Μια χαρά ήταν η συνεργασία. όλη την Ευρώπη και με, το Ισραήλ συνεργαζόμαστε. Σα είπα, καμιά εκατοστή προγράμματα έχουμε τρέξει. Τέλο. Πώς θα έχουμε κάποια εφαρμογή που να διακρίνεται από ισορροπία. Εδώ είναι πολιτική απόφαση για το πώς θα γίνει η κατανομή η γεωγραφική. Και πώς θα υπάρχουν εγγύσεις συμμετοχής αρκετών χωρών για κάθε πρόγραμμα. Για την υλοποίηση των προγραμμάτων. Όμω θα πρέπει να υπάρχει εξειδίκευση τη κάθε περιοχής στην Ευρώπη, ούτω ώστε να μην ασχολούνται όλοι με όλα. θα πρέπει ίσως να δανειστούμε ιδέες από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος για ε, ε, αυτό που έχουν εκεί που το λένε prime contractors και πρώτοι για κάποιες μεγάλες βιομηχανίες που ασχολούνται με τα του διαστήματος προοικοδοτούνται ενισχύονται αυτές οι βιομηχανίες, αλλά οφείλουν να συνεργαστούν με μικρότερες βιομηχανίες, με υπεργολάβους ας πούμε. Ίσως αυτό θα ήταν μια λύση και για μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στόμα. <clears throat> Θα αρχίσω με τα σχόλια του κυρίου Έλερ. Γερμανικά όμως να τα πω για τα θέματα της αριστείας. Αν ορίζεται αυτό εθνικά ή όχι. Για το Ινστιτούτο Φράνχοφερ μπορώ να σας πω ορίζεται, διότι υπάρχουν ε, Ινστιτούτα και Ιδρύματα που δεν κάνουν καθόλου στρατιωτική έρευνα και κάποια άλλα που κάνουν. Δεν υπάρχει διάκριση. Δεν υπάρχει κανένας που να έρχεται και να λέει ότι εγώ κάνω στρατιωτική έρευνα, δεν μπορώ να κάνω δημοσιεύσεις, δεν μπορώ να το δικαιολογώ, όχι, δεν υπάρχει λόγος που να εξαιρείσαι και να θεωρείς ότι είσαι άριστος χωρίς έλεγχο. Και έχουν παρέλθει οι καιροί εκείνοι που ενισχύαμε οικονομικά κάποιο Ινστιτούτο που είχε πρόβλημα γιατί δεν πάει καλά. Αυτά έχουν τελειώσει. Ε, συνεργαζόμαστε με τις ΗΠΑ με τη Γαλλία, με το Ισραήλ. Πάντα όλα αυτά τα προγράμματα ε, είναι μετά από διακυβερνητικές συμφωνίες για κοινά ερευνητικά προγράμματα. Αυτή τη στιγμή έχουμε προσωπία του Ινστιτούτου Φράνχοφερ στο Ισραήλ για συζήτηση θεμάτων αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Υπάρχουν πάρα πολλοί σαφείς κανόνες λοιπόν για το πώς ε, ρίζεται η αριστεία και διεθνώς εθνόση συνεργασία ε, είναι δυστυχώς με οι Ηνωμένε Πολιτείε, Ισραήλ και Γαλλία. Για τη συνεργασία είπατε αν έχει πρόβλημα. Ε, μέχρι τώρα ε, είναι διακυβερνητικές μόνο οι συνεργασίες με το Ισραήλ ή με ε, τη Γαλλία. Μέχρι τώρα πάντα υπάρχει κάποιος εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Εγώ θα επιθυμούσα στην έρευνα για την ασφάλεια να μπορούν να εργάζονται ανεξάρτητα οι ερευνητές. Γιατί πάντα χάνουμε χρόνο μέχρι να συμφωνήσουν οι κυβερνήσεις. Ε, πρέπει να αλλάξει αυτό ε, και στον αμυντικό και στον πολιτικό τομέα. Στη συνέχεια έγινε μια ερώτηση από την κυρία Λόζινγκ για την ομάδα προσωπικότητων. Έχετε δίκιο. Ε, θα πρέπει όμως από κάπου να ξεκινήσουμε. Έτσι προέκυψε αυτή η ομάδα προσωπικότητων ε, με βάση την παγκόσμια στρατηγική. Από εκεί θα πρέπει να αρχίσετε την κριτική σας. Και όταν διάβασα αυτή την ε, στρατηγική είπα, μα τι φιλόδοξοι είναι οι άνθρωποι. Πώς θα φτάσουμε σε αυτή την παγκόσμια στρατηγική για να γίνει αυτό, χρειάζονται να γίνουν κάποια πράγματα όμως. Βλέπω όμως ε, μεγάλη αντιστοιχεία Ε, τα τελευταία δέκα χρόνια ακολουθήσαμε την ίδια πορεία για την έρευνα. Εχθές ήμουν ε, στη συζήτηση εδώ στις Βρυξέλλες με το Υπουργείο Έρευνας. Αρχίσαμε με τις τεχνολογίες, αναπτύξαμε κάποιες ιδέες, αλλά μας είπαν ναι, αλλά τώρα κάτι μας λείπει. Ε, λείπουν οι κοινωνικοί επιστήμοντες, λείπουν οι νομικοί, οι καθηγητές διεντολογίας, ηθικής, όλοι αυτοί θα πρέπει να συμμετέχουν στην Επιτροπή Προσωπικότητων, βεβαίως άκουσα ότι θα υπάρξει και δεύτερη ομάδα προσωπικότητων, γιατί όχι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Καλό είναι πάντα να ακούγονται και άλλες φωνές. Ας πούμε, ε, στην έρευνα για την πολιτική ασφάλεια, στο μεταξύ είναι υποχρέωση για κάθε έργο να υπάρχει ανάλυση ηθικής και διοντολογίας με ερωτηματολόγιο. Δεν έχω κανένα πρόβλημα, θα μπορούσαμε και για τα αμυντικά ερευνητικά προγράμματα να το κάνουμε. Έχουν γίνει κάποιες πρώτες προσπάθειες. Γιατί υπάρχουν ε, κάποια πράγματα που αποκλείονται, α πούμε, για τα μέσα μαζικής καταστροφής. Αυτό αυτά όλα είναι σε εξέλιξη. Ε, στην έρευνα ασφαλείας ε, την τελευταία δεκαετία έχουν γίνει προσπάθειες. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να διευρυνθεί η ομάδα προσωπικότητων και να συμπεριληφθούν και άλλα στοιχεία νομικά, κοινωνικά, ηθικής και δεδολογίας. Στη συνέχεια, ο Πολωνός εκπρόσωπος ρώτησε ε, για το Ινστιτούτο Φρανχόφερ στη Γερμανία και είδε το χάρτη της χώρας. Πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα έχετε, αλλά σε μερικά κρατήδια έχουμε μικρότερη εκπροσώπηση. Για ποιο λόγο? Πας σε ένα καθηγητή και του λες θέλεις να στήσεις ένα Ινστιτούτο ε, στο τάδε κρατήδιο και όταν χρειάζεται να αυτοχρηματοδοτηθεί, να ξεκινήσει από το μηδέν μια προσπάθεια, ε, υπάρχουν κάποια κρατήδια που δεν έχουν πολύ μεγάλη βιομηχανική ανάπτυξη και δεν τα προτιμούν. Ε, βγαίνουν στα κρατήδια που υπάρχουν ήδη στημένες βιομηχανίες και έχουν εταίρους. Πάντως είναι σημαντικό αυτό που είπατε. Αλλά προσπάθειες γίνονται και στην Ανατολική Γερμανία. όταν ενώθηκε η Γερμανία, Μα ανέθεσε η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση στο Ινστιτούτο Φρανχόφερ να αναλύσουμε τα Ινστιτούτα της Ακαδημίας Επιστημών της Ανατολικής Γερμανίας και να αποφασίσουμε αν θα τα κλείσουμε ή αν θα τα μεταξελίξουμε σε τμήματα του Ινστιτούτου Φρανχόφερ. Πριν από λίγο γιορτάσαμε τα 20 χρόνια την επέτειο ένταξης των Ανατολικών Ινστιτούτων. Όλοι είναι πάρα πολύ επιτυχείς μετά από 10 χρόνια το κατάφεραν γιατί είχαν έκτακτες ρυθμίσεις μια δεκαετία να φτάσουν και να ακολουθούν τους ίδιους κανόνες και τα ίδια πρότυπα με τα Ινστιτούτα που από καιρό και πολλές δεκαετίες λειτουργούν στη Δυτική Γερμανία. Και έχουμε ιστορία επιτυχίας τώρα ότι στήσαμε Ινστιτούτα Φρανχόφερ και στην προενατολική Γερμανία. Αλλά τι χρειάζεται, 10 χρόνια μαζική χρηματοδότηση από το κράτος και ε, λίγη από τα ευρωπαϊκά κονδύλια διαρθωτικά ταμεία, αλλά θα πρέπει να πούμε ότι έτσι έχει ζωή. Υπάρχουν και φάροι, δρέσδι, γένα, λειψία ενδεχομένω. Τώρα δεν μπορείς να περιμένεις σε κάθε επαρχία της πρώην Ανατολικής Γερμανίας να έχουμε την ίδια υποδομή και την ίδια έρευνα και δικτύωση. Υπάρχουν μεν και κάποιες φωτεινές εξαιρέσεις Μια ερώτηση που έρχεται συχνά είναι το χάσμα μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένων Πολιτειών. Ισχύει αυτό. Όχι σε όλους τους τομείς, σε μερικούς. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπου η Γερμανία, η Ευρώπη είναι ηγέτες, ας πούμε, οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αντιγράψουν το δικό μας μοντέλο του Φραουνχόφερ, δεν το έχουν μέχρι στιγμή στη βιομηχανία τους. Ας πούμε, γίνεται και η παραγωγή στον πολιτικό τομέα έχουμε παραγωγή, αλλά στο στρατιωτικό υπολοιπόμαστε και έχουμε και καθυστέρηση. Και φυσικά όταν έχουν πενταπλάσια χρηματοδότηση στις ΗΠΑ θα έχουν τουλάχιστον διπλάσια απόδοση. Για τα προβλήματα των εξαγωγών, απάντησε ο συνάδελφος του Βιλμάνιε για το θέμα της συνεργασίας με την Ανατολική Ευρώπη στο Ινστιτούτο Φρανχόφερ. Το προσπαθούμε, αλλά αυτή τη στιγμή αυτή η υπόθεση. Είναι αρκετά μικρή η συνεργασία μας. Επίσης ρωτήσατε τι γίνεται με τις ανισορροπίες. Ανισορροπίες θα υπάρχουν πάντα. Γιατί σας είπα υπάρχουν φωτεινές εξαιρέσεις, κάποιοι φάε, ε, ανακρατήδιο μπορεί να είναι ένας ή δύο, αλλά θα πρέπει εκεί να επικεντρωθούμε όπου εξειδικεύεται κάποιος κλάδος της ε, βιομηχανίας. Κάποιος ρώτησε μήπως έχουμε υπερβολικές φιλοδοξίες, μήπως να αρχίσουμε από μικρά έργα. Εγώ θα απαντούσα. Ας κάνουμε το ίδιο που κάναμε με την έρευνα ασφαλείας. Έχουμε τέσσερις κατηγορίες έργων εκεί, μικρά και με μικρούς εταίρους που συμμετείχαν πραγματικά για θέματα θεμελιώδη μέχρι και μεγάλα ε, προγράμματα ε, ε, επίδειξης πανευρωπαϊκά. Ο κύριος Έλερ αναφέρθηκε στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια που θα έπρεπε ε, να ελέγξουν, να δοκιμάσουν συστήματα ασφαλείας ενία Ξέρω εγώ Αθήνα, Παρίσι και άλλα αεροδρόμια. Αναφερθήκατε σε ένα διπλωμάτη για τη στρατηγική αυτονομία. Ε, είπε ότι είναι ανέφικτη. Δεν είναι ανέφικτη, είναι εφικτή. Χρειαζόμαστε στρατηγική αυτονομία. Ορισμένοι την ονομάζουν μη εξάρτηση. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Ε, για τη διαστημική υπηρεσία. Αν θέλει μια ευρωπαϊκή εταιρεία να φτιάξει ένα δορυφόρο και θέλουν να πάρουν ε, ανταλλακτικά από τις Ηνωμένε Πολιτείε που είναι στη λίστα του ΙΤΑΡ του κανονισμού για το Διεθνές Εμπόριο Όπλων πρέπει να στείλουμε όλο το σχέδιο στις Ηνωμένες Πολιτείες προς έγκριση κτλ. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή πούμε για τους πυράβλους κρούς κάποιος αγόραζε τα τελευταία δέκα χρόνια και κάποια στιγμή ήρθε μια επιστολή, σταματάμε να σας πουλάμε πυράβλους. Για ποιο λόγο, γιατί θα πρέπει να κάνετε πλήρη αναφορά και εξήγηση τι τους θέλετε, πού θα τους χρησιμοποιήσετε κτλ. Και η γερμανική κυβέρνηση ότι καλά θα δούμε να φτιάξουμε δικούς μας. Ε, η στρατηγική αυτονομία είναι κάτι που πρέπει να συζητήσουμε σε λεπτομέρειες. Ε, ε, σήμερα η βιομηχανία χρησιμοποιούν όλοι εξαρτήματα από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά είπα, αν είναι στον κατάλογο ε, ΆΙΤΑ, πρέπει κάθε φορά να κάνουμε επιστολές, δικαιολογία, τι το θέλουμε, πού θα το πάμε, πού θα το εξάγουμε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ. Thank you very much. Ευχαριστούμε πολύ και τους τρεις εμπειρογνώμονές μας και έτσι εδώ ολοκληρώνεται αυτό το σημείο στην εμερήσια διάταξη και θα περάσουμε ευθύ αμέσως στο επόμενο σημείο που είναι οι εξελίξεις στην κατάσταση ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Ευχαριστούμε πολύ.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 Ladies Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Αρχίζουμε ευθύ αμέσω. Το επόμενο σημείο στην ημερήσια διάταξη, όπω είπαμε, είναι οι εξελίξει στην κατάσταση ασφάλεια στη Μέση Ανατολή. Πολύ επίκαιρο το θέμα και πολύ σημαντικό βέβαια. Πρέπει να σας ενημερώσω ότι ένας από τους εξέχοντες προσκεκλημένους μας δεν μπόρεσε τελικά να έρθει. Κάτι έκτακτο συνέβη στο Παρίσι. Η κυρία Φλωράν Σκάουπ, δηλαδή αναπληρωτής διευθυντής του Ινστιτούτου Μελετών Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν θα έρθει να μας κάνει την παρουσίασή σα. Η γραμματεία ίσως θα μπορούσε να τη ζητήσει να μας στείλει ε, γραπτά ό,τι είχε ετοιμάσει. ώστε να ενημερωθούμε μια που τη έτυχε αυτό το εκτακτό και δεν μπόρεσε να έρθει. Κάποια καταστροφή τη συνέβη. στο σταθμό στο Παρίσι και δεν μπόρεσε να έρθει. Οπότε θα ακούσουμε τους άλλους δύο εμπειρογνώμονες. Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω εδώ τον κύριο Νουίτζι Ναρμπόνε που είναι ανώτερο σύμβουλος για την Μέση Ανατολή και την Βόρεια Αφρική στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και την κυρία Κριστίνα Κάους, η οποία είναι ανώτερη ερευνήτρια στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ των Ηνωμένων Πολιτειών. Νομίζω ότι όλοι γνωρίζουμε πώς έχει η κατάσταση και ευχαρίστω να ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες για τα διέξοδα και για τις ενδεχόμενες λύσεις. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, είναι πολύ επίκαιρη η σημερινή συζήτηση. Φαίνεται ότι συνεχώς έχουμε νέα γεγονότα στην Μέση Ανατολή και κάποια από αυτά τουλάχιστον επηρεάζουν ολόκληρη την περιοχή. Οπότε θα προσπαθήσω εδώ να εξετάσω μαζί σας τα σοβαρά γεγονότα των τελευταίων εβδομάδων και αυτό υπό το φως των εντάσεων που μπορεί αυτά να προκαλέσουν, όπως επίσης θα εξετάσω και ποιοι είναι οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μειώσει ακριβώς τις εντάσεις και να αποκλιμακώσει την ε, σύγκρουση στην περιοχή. Επίσης, λαμβάνω υπόψη μου ότι υπάρχουν και στρατηγικές συμμαχίες, ότι υπάρχουν γρήγορες πολιτικές και άλλες εξελίξεις Έχουμε να κάνουμε με μια ε, περιοχή η οποία έχει αποσταθεροποιηθεί πάρα πολύ από συνεχόμενες κρίσεις και σίγουρα δεν χρειάζεται παρετέρω αποσταθεροποίηση. Συνεπώς, θα προχωρήσω στην ανάλυση μου εξετάζοντας τα διάφορα γεγονότα και θα σας πω τι συμβαίνει στις διάφορες χώρες, στα διάφορα πεδία και ποιες είναι οι επιπτώσεις των γεγονότων αυτών και τι σχεδιάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση σε αυτά. Και θα αρχίσω με τη Σαουδική Αραβία, όπου βέβαια έχουμε σημαντικές εξελίξεις. Πρώτα απ' όλα ήδη α, στις γενιές που βρίσκονται επικεφαλής στη Σαουδική Αραβία ε, περνάμε από μια παραδοσιακή ε, συνένεση στην λήψη αποφάσεων. Ο Μοχάμεντ Μπιλατσμάν, ο πρίγκιπας, ανέλαβε την ευθύνη για διάφορα θέματα κλειδί οικονομικά και στρατιωτικά συστήματα, ε, προχώρησε σε μεταρρυθμίσεις και σχεδιάζει και άλλες μεταρρυθμίσεις που θα αλλάξουν σίγουρα ε, την όψη της χώρας, προσπαθώντας να διαφοροποιήσει την οικονομία της χώρας απομακρυνόμενος από τον άνθρακα και έχοντας υπόψη τον ορίζοντα 2030. Ε, κάνει αλλαγέ, όπω για παράδειγμα επιτρέπει στι γυναίκε να οδηγούν, να συμμετέχουν σε δημόσιε εκδηλώσει. Και επίση, στα πλαίσια αυτά, ξεκίνησε και μια εκστρατεία κατά τη διαφθορά, η οποία έχει ω ε, στόχο ε, διάφορε σημαντικές προσωπικότητες επιχειρηματικέ στο Βασίλειο. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Οι αλλαγές τώρα στο εσωτερικό συνδυάζονται και με επιθετικές κατά κάποιο τρόπο δράσεις και ρητορική της Σαουδικής Αραβίας στην περιοχή, κατά του Ιράν, για παράδειγμα. Στην Ιεμένη είχαμε τον πύραυλο κατά της Ιεμένης, κάτι απαράδεκτο, και υπάρχει κίνδυνος παρετέρω επιδίνωσης της κατάστασης στην περιοχή. Η Συμμαχία συνεχίζει τους βομβαρδισμούς ε, από αέρα. Ε, προσπαθεί να αποφύγει βέβαια στον άμαχο πληθυσμό καταστροφές και θανάτους. Έπειτα υπάρχουν ε, και τζιχαστικές τρομοκρατικές οργανώσεις οι οποίες παγιώνουν τη δύναμή τους. Η Εμένη είναι η χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο και η κρίση κινδυνεύει να επιδεινώσει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Η διαδικασία των Ηνωμένων Εθνών δεν έχει οδηγήσει σε σημαντικά αποτελέσματα προς το παρόν και φαίνεται ότι υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια για διπλωματική δράση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να φτάσει σε όλες τις πλευρές και να πετύχει κάποιο πολιτικό διάλογο. Εκ παραλλήλου είχαμε και την κρίση στο Κατάρ που άρχισε τον Ιούνιο και εξακολουθεί να παραμένει, εμποδίζει το έργο μας και δημιουργεί βέβαια εντάσεις γύρω από την περιοχή του κόλπου. Παρετήθηκε επίσης ο Πρωθυπουργό Χαρίρη του Λιβάνου και πήγε στο Ριάτ, κάτι το οποίο μας προβληματίζει όσον αφορά τη σταθερότητα στο Λίβανο. Υπάρχουν ανησυχίες για το πολιτικό μέλλον του Λιβάνου και υπάρχει κίνδυνος τα γεγονότα αυτά να υπονομεύσουν τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα, τους τελευταίους μήνες τουλάχιστον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από τα δικιά της την πλευρά εξακολουθεί να στηρίζει το διάλογο για να λυθεί η θεσμική αυτή κρίση και προσπαθεί να διασφαλίσει να γίνουν κοινοβουλευτικέ εκλογές την Άνοιξη όπως προβλέπεται προς το παρόν. Για το Ιράν, η Ευρωπαϊκή Ένωση θεωρεί ότι η διατήρηση και η συνεχής εφαρμογή της συμφωνίας GPC με το Ιράν, την οποία εγγυάται η Αντιπρόεδρος κυρία Μογκερίνη, έχει τεράστια σημασία. Συγχρόνως μας απασχολούν και άλλα ζητήματα. Το θέμα της ικανότητας της πυρηνικής, των πυράβλων, τι ρόλο παίζει το Ιράν. Και είναι πράγματα τα οποία βεβαίως και συζητούμε πάντα κάθε φορά που έχουμε διάλογο. Προσπαθούμε να προοδεύσουμε σε αυτά τα ζητήματα όσον αφορά τις σχέσεις μας με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, παρά τα προβλήματα στην περιοχή, κάνει έκκληση για διάλογο και ηρεμία. Αποκλιμάκωση και απομάκρυνση από την πόλωση και τον κατακαιρματισμό στην περιοχή. Κάτι το οποίο βέβαια είναι και εν μέρη αιτία της ε, κρίσης στην περιοχή και της σύγκρουσης που έχουμε τα τελευταία χρόνια. Συνεχίζω τώρα με άλλα πεδία. Ιράκ, η πολιτική κατάσταση στο Ιράκ. Έχουμε εκεί κάπως πιο ενθαρρυντικές εξελίξεις. Υπάρχει μια προσέγγιση του Ιράκ με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου. Κάτι πολύ ενδιαφέρον. Θετικό επίσης είναι και ο τρόπος με τον οποίο η Ιρακινή κυβέρνηση και της περιοχής αντιμετωπίζουν την κρίση μετά το δημοψήφισμα. Εμείς δουλεύουμε πάνω σε μια νέα στρατηγική Ιράν-Ιράκ που θα είναι έτοιμη στις αρχές του 2018 και είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε το Ιράκ για μια σταθερότητα και συμφιλίωση στη χώρα. Το Ιράκ πρέπει να απομακρυνθεί από τον κατακαιρματισμό μεταξύ των διαφόρων φυλών που αποτέλεσε πρόβλημα τα τελευταία χρόνια και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζει και τη διαδικασία νοικοδόμησης. Πολύ σημαντικό και τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις επίσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, προσπαθεί να έχει μία αποστολή άμυνας και ασφάλειας προκειμένου να βοηθήσει. Στη Συρία το ΝΤΑΣ ελέγχει τώρα λιγότερο από 5%. Έχουμε πετύχει εκεί κάποια βελτίωση. Παραμένουν όμως φοβερές ανησυχίες όσον αφορά τη διακυβέρνηση και την βοήθεια στις περιοχές που έχουν απελευθερωθεί από την ΤΑΕΣ, από την ISIS. Και φυσικά πάντα θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις αιτίε που οδήγησαν στην άνοδο του ISIS και που οδήγησαν και στην τζιχαντιστική τρομοκρατία. Δεν υπάρχει σαφής πρόοδος όσον αφορά την αποκλιμάκωση στη Συρία και εξακολουθούν να γίνονται βομβαρδισμοί από αέρος από την Ρωσία και από άλλους παίκτες στην περιοχή, σε κάποιες περιοχές. Ε, κάτι βέβαια που οδηγεί σε δίνει τον άμαχο πληθυσμό και ανθρωπιστική βοήθεια προκειμένου να φτάσει δεν τα καταφέρνει. Παρ' όλα αυτά η πολιτική βούληση για επίλυση ε, παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Θέλουμε να φτάσουμε σε διαπραγματεύσεις για να υπάρξει ενότητα στη Συρία, να μην υπάρξει κατακαιρματισμός και να μπορέσουν να επιστρέψουν με ασφάλεια οι πρόσφυγες. Υπάρχει διαδικασία των Βρυξελών από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον διάλογο αυτό και προσπαθούμε να δούμε και αν τα 9,5 εκατομμύρια τελικά φτάνουν, δισεκατομμύρια, δεν φτάνουν στον προορισμό τους, έτσι όπως αποφασίστηκε πέρυσι μάλλον φέτο στην διάσκεψη των Βρυξελών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τη διαδικασία και χρησιμοποιεί ό,τι μέσα μπορεί προκειμένου να προχωρήσουμε σε μια νέα διάσκεψη ε, Βρυξελών τον Μάιο του 2018. Όσον αφορά την ειρηνευτική διακασία στη Μέση Ανατολή, η βία παραμένει παρούσα ήδη από το 2015 και μετά, η ειρηνευτική διαδικασία παρόλα αυτά παραμένει ζωντανή σε, ε, σε επίπεδα όμως που δεν εξελίσσεται, παραμένει δηλαδή στάσιμη και οι Παλαιστινιακές αρχές πρέπει να αναλάβουν τις ευθύνες τους από 1η Δεκεμβρίου στη Λωρίδα της Γάζας, γιατί είχαμε και αυτή την εξέλιξη όσον αφορά την Γάζα και εμείς στηρίζουμε την Παλαιστινιακή Αρχή προκειμένου να αναλάβει τον πλήρη έλεγχο στην ε, περιοχή. Φυσικά υπάρχουν πολλές δυσκολίες, ο φοπλισμός της Χαμάς για παράδειγμα, κάτι το οποίο ζητούν και το Ισραήλ και η Παλαιστινιακή Αρχή. Τώρα ο πρόεδρος της Αιγύπτου, Αλ Σίση. Ε, και εδώ έχουμε την ενευτική διαδικασία που στηρίζεται και από τον Αραβικό Σύνδεσμο και έτσι ελπίζουμε να υπάρξει κάποια εξέλιξη στην ενευτική διαδικασία εκεί. Οι διεθνείς παράγοντες καλωσορίζουν την δέσμευση των ενδιαφερομένων πλευρών και βλέπουν την ειρηνευτική αυτή πρωτοβουλία σαν μια δυνατότητα να δημιουργηθεί μια νέα δυναμική και νέα κίνητρα για ειρήνευση. Επιπλέον, οι Ηνωμένε Πολιτείες δηλώνουν έτοιμες να αναπτύξουν νέα αποστολή Χιούμπαμ Ράφα. Τέλος, στη Λιβύη. Η κατάσταση παραμένει ρευστή. Η Λιβύη βέβαια δεν αποτελεί μέρος της Μέση Ανατολής αυτής καθ' αυτής, παρόλα αυτά συνδέεται με τις συγκρούσεις στην περιοχή. Η κατάσταση εκεί παραμένει ρευστή λοιπόν, υπάρχει ελάχιστη πρόοδος οικονομικά, ο πολιτικός διάλογος, σύνταγμα, όλα αυτά προχωρούν αργά και η κατάσταση ασφάλειας είναι μεν κάπως ήρεμη παρόλο που σποραδικά υπάρχει βία. παραμένουν δυσκολίες για βελτίωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κατάστασης και για την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων. Η προσπάθεια όμως παραμένει, συνεχίζεται. Σποραδικά σε διάφορες περιοχές, Βεγάζη, Μπέν και αλλού, ε, υπάρχουν κάποιες εκδηλώσεις βίας. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά και στηρίζει τις προσπάθειες του ΟΗΕ και είναι έτοιμη να συνεισφέρει για θέματα δικαίου, στις αποστολές BAM για παράδειγμα και στην οικονομική στήριξη για μεταρρυθμίσεις. Στηρίζουμε για NSRG το σχετικό πρόγραμμα και ελπίζουμε να μπορέσουμε και εμείς να συνεισφέρουμε για την βελτίωση στη Λιβύη. Αυτή είναι η εικόνα. Τελειώνοντας, μπορώ να πω ότι η κλιμάκωση δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει κάθε άλλο, ούτε στο Ιράκ, ούτε στη Ιεμένη, ούτε πουθενά, ούτε ε, οι πύραυλοι που εκτοξεύονται. Οπότε χρειάζεται μια λύση διαρκεία, σήμερα περισσότερο από ποτέ. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας σε πολλά από αυτά τα τόσο λεπτά μέτωπα. Ευχαριστώ. Θα παρακαλέσω τώρα την κυρία Κριστίνα Κάους, ανώτερη ερευνήτρια στο Γερμανικό Ταμείο Μάρσαλ των Πολιτειών, να λάβει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, που με καλέσατε ε, σε αυτή τη συνεδρίαση. Θα ήθελα να αναφερθώ σε τρία βασικά θέματα. Από εκεί που σταμάτησε ο κύριος Ναρμπόνε να συνεχίσω την ευρύτερη εικόνα και μετά να σταθώ σε κάποια σημεία που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή τις επόμενες εβδομάδες και μήνες ως αποσταθεροποίηση και σύγκρουση. Δεύτερο, το ρόλο της ε, κυβέρνησης Τραμπ και στον υπόλοιπο χρόνο μου θα μιλήσω λίγο για το λόγο ε, ε, του κυβερνοχώρου στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Ε, έχουμε ανακατατάξεις και κλιμακώσεις ε, τελευταία βρισκόμαστε σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο. Οποιαδήποτε παρουσίαση για τις συγκρούσεις ε, στη Μέση Ανατολή λέει ότι είμαστε σε παραμονές έκρηξης κάθε φορά όποιος αναφέρεται σε αυτά. Αλλά σήμερα πραγματικά υπάρχει κίνδυνος. Αν δούμε το status quo για μείζωνα έκρηξη μάλιστα στο τρίγωνο μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Ιράν και Ισραήλ. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι που το θετούν αυτό. Ένας από αυτούς είναι η πρόσφατη συμμαχία Σαουδικής Αραβίας Ισραήλ με την υποστήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών που επέλεξε να διαλέξει πλευρά σε αυτή την πόλωση της περιοχής. Και το επίκεντρο είναι αυτό το τρίγωνο οι βασικές ε, εξελίξεις που θα πρέπει να παρακολουθούμε το επόμενο διάστημα δύο-τρεις εβδομάδες είναι η κρίση στο Λίβανο μετά τις συζητήσεις που γίνονται στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών μήπως ε, επιπληθούν και πάλι κυρώσεις στο Ιράν και αυτό να επεκταθεί και στη Χεσμολάχ και πώς θα αντιδράσει το Ιράν, πώς μπορεί να αντιδράσει το Ισραήλ και αν αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μια πολιτική κρίση στο Λίβανο. Η ήδη σοβούσα πολιτική κρίση στο Λίβανο, μήπως μπορεί να γίνει τελικά στρατιωτική σύραξη, γιατί υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο. Ο αποκλεισμό της Ιεμένης που ανέφερε και ο κύριος Ναρμπόνε δεν μπορεί να Ε, υπερτιμηθεί. Δεν, δεν ξέρω τι εννοείτε κύριε Ναρμπόνε. Δεν θυμάμαι την ακριβή διατύπωσή σας. Είπατε ότι δεν υπάρχει χώρος για περαιτέρω διπλωματική πίεση στη Σαουδική Αραβία. Χρειάζεται. Ε, οπωσδήποτε για να αφήνει τη βοήθεια να περνά προς την Ιεμένη. Είναι μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, μεγαλύτερη ε, δεκαετιών χολέρα, λοιμός. Αρχίζει ο κόσμος και τα παιδιά να πεθαίνουν από την πείνα στην πιο φτωχή αραβική χώρα. Τις επόμενες εβδομάδες και μήνες θα πεθάνουν εκατομμύρια άνθρωποι. Εάν δεν υπάρξει πλήρης ε, πρόσβαση στα λιμάνια. Και έγινε έρευνα από τον ΟΗΕ ε, και τα, οι ε, εφοδιοπομπές εκεί δεν ε, μεταφέρουν πυράβλους και όπλα. Ίσα ίσα η Σαουδική Αραβία και μένα χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα και να χρησιμοποιήσει ως όπλο τις ασθένειες και το λοιμό. Αλλά ας μην λησμονούμε ότι είναι παιδί του Μοχάμετ Μπιν Σάλμαν η Εμένη ο οποίος θα πρέπει να κερδίσει αυτό τον πόλεμο για να εδρεώσει και την ίδια του τη φήμη και το κύρος του μέσα στη Σαουδική Αραβία. Υπάρχει μέγας χώρος λοιπόν για πίεση στη Σαουδική Αραβία να σταματήσει και να αφήσει την πλήρη πρόσβαση προ τους λιμένες και μεταξύ αυτών εκείνων που ελέγχουν. Δεν χρειάζεται να είναι πλήρης ο αποκλεισμός, μπορούν να ελέγχουν τις νεοπομπές, ό,τι θέλουν τα καράβια. Είναι τελείως άχρηστο αυτό να διακινδυνεύουν να χάσουν τη ζωή τους εκατομμύρια ανθρώπων. Για το Λίβανο. Όπως είπα και προηγουμένως, εάν το Κογκρέσο, και αυτό δεν έχει διευκρινιστεί καθόλου, ε, αποφασίσει οι κυρώσεις να επεκταθούν και στη Χεσμολά, κάτι θα προκαλέσει κάποια αντίδραση. Είχε πολλά που τη στηρίζει το Ιράν. Αλλά στο Λίβανο αυτό μπορεί να οδηγήσει μια, σε μια κατάσταση όπου επιτέλους θα έχει μια ε, πρόφαση το Ισραήλ για να επέμβει, ε, να παρέμβει στρατιωτικά μαζικά κατά της Χεσμολά στο Λίβανο. Ουσιαστικά αυτό σημαίνει πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Άρα αν κάνουμε ένα βήμα πίσω και δούμε ολόκληρη τη σύγκρουση Σαουδικής Αραβίας-Ιράν, η Σαουδική Αραβία έχει πολύ καλούς λόγους να μην είναι ευχαριστημένη με την επεκτατική στρατηγική του Ιράν. Ταυτόχρονα όμως είναι σε σαφές μειονέκτημα η Σαουδική Αραβία. Θα ήθελα λίγο να σας δώσω αυτή την εικόνα ε, του πληγωμένου θηρίου, του λιονταριού που χυμάει ανεξέλεκτα σε όλους. Υπάρχει μια άτυπη συμμαχία τώρα Αραβία σε Ισραήλ που μπορεί να οδηγήσει σε κλιμάκωση. Ταυτόχρονα η Σαουδική Αραβία δεν μπορεί να κάνει πολλά πράγματα εναντίον του Ιράν. Τους αντιπροσώπους μπορεί να έχει ως ε, εχθρούς και να επιτίθεται ε, ας πούμε στη Συρία και ε, ίσως μεθαύριο στο Λίβανο αλλά αυτό λύνει προβλήματα, αλλά δημιουργεί άλλα τόσα για τη Σαουδική Αραβία. Δεν είναι στρατηγική μακροχρόνια. Και στο παρελθόν χειραγώγησε την πετρελαϊκή κρίση και τη χρησιμοποίηση. Ε, αλλά δεν μπορεί να το κάνει πια, ούτε να το επομιστεί οικονομικά, γιατί τα οικονομικά της χώρας δεν είναι και σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Άρα, ο μόνος τρόπος ε, να σταματήσει αυτή η κλιμάκωση είναι η Σαουδική Αραβία και το Ιράν με κάποιο τρόπο να κάνουν κάποιο διάλογο, έστω και άτυπο. Δεν πρόκειται το Ιράν να υποχωρήσει και η Σαουδική Αραβία δεν έχει συμφέρον και δεν είναι προς το συμφέρον καθενός να εκραγεί ολόκληρη η περιοχή εκεί. Ανταυτού, με τη στήριξη των ΗΠΑ η Σαουδική Αραβία επιδιώκει να στριμώξει το Ιράν στη διεθνή απομόνωση. Να το εξωθήσει προς τα εκεί και εκεί η Ευρώπη θα πρέπει να αντιταχθεί. Επίσης, η προσέγγιση με το Ισραήλ είναι μια στρατηγική κίνηση για να φτιάξουμε μέτωπο κατά της Τεχεράνης, με τη σιωπηρή ε, ευλογία των Ηνωμένων Πολιτειών. Εμείς θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε ε, τη συμφωνία με το Ιράν για να αποκλιματιθεί η κατάσταση και στο Κατάρ και σε άλλες περιοχές γύρω από τη Σαουδική Αραβία και να δημιουργηθούν διάλογοι, διάβλη μάλλον επικοινωνίας Ιράν-Σαουδικής Αραβίας. Έρχομαι στο ρόλο της κυβέρνησης Τραμπ σε όλα αυτά, που πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία. Όχι μόνο στη Μέση Ανατολή, γενικότερα. Μέχρι τώρα έχουμε πλήρως παρατηρήσει ε, το, τη στάση, αυτή τη ρητορική ε, που είναι παρορμητική και παμφωτερίζουσα. Ποια είναι η βασική αλλαγή τώρα στην κυβέρνηση Τραμπ. Ε, αυτή η σύγκρουση με το Ιράν. Ακόμα και αν είναι ρητορική αυτή η έξαρση, η αποχώρηση από τη συμφωνία, ακόμα και αν δεν καταλήξει σε τερματισμό της ή σε κατάργησή της, στέλνει κάποια μηνύματα από μόνη της. Ένα μήνυμα σύγκρουσης με το Ιράν, έτσι κι αλλιώς που έχει περιδοτήσει σειρά αντίδρασεων, ας πούμε, εχθρικών. Και στέλνει και ένα μήνυμα και προς άλλους ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε δεν τηρούν τις συμφωνίες, δεν τιμούν τις συμφωνίες που έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση. Και εδώ σκέφτομαι και τη Βόρεια Κορέα. Το να επιλέξεις με ποιον είσαι σε αυτή την περιφερειακή σύγκρουση έρχεται σε κατάφορη αντίφαση με την πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή την τελευταία δεκαετία. Ότι προσπαθούσαν λογικά να τηρήσουν ίσες αποστάσεις, ισορροπία δυνάμεων, ταυτόχρονα συνομιλώντας με όλους. Και χωρίς να ευνοούν μια χώρα. Τώρα τι κάνουν ή τι φαίνεται ότι κάνουν. Το αντίθετο επιλέγουν ότι είναι με τη συμμαχία του Ισραήλ με τη Σαουδική Αραβία κατά του Ιράν. Και αυτό είναι πάρα πολύ επιβλαβές, γιατί αμφιβάλλω πάρα πολύ κατά πόσο η Σαουδική Αραβία θα, προχωρήσει, ή θα προχωρούσε τόσο πολύ αν δεν είχε τις ιοπηρές ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ηρωνικό. Αλλά αν βγάλουμε το Ισλαμικό κράτος από την εικόνα, από το κάδρο αυτό, τώρα η προτεραιότητα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν σημαίνει ότι έχει αλλάξει επειδή κατατροπώθηκε το Ισλαμικό κράτος και είναι ε, ηρωνικό αυτό. Τώρα που χάθηκε το Ισλαμικό κράτος μπορεί να στοχεύσει το Ιράν, που, έχει, που είναι η μόνη χώρα που έχει κάποιο σχέδιο για την περιοχή και θα επωφεληθεί από το τέλος το ISIS, βασικά το Ιράν. Δεν ξέρω, κύριε Ναρμπόνε, θα μπορούσατε να το σχολιάσετε κι εσείς για το που βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, σε σχέση με τη συμφωνία με το Ιράν και τα όσα συζητεί το Κογκρέσο. Μάλλον θα συγκρουστεί η Ευρώπη ε, με το Κογκρέσο λόγω της δικής του συγκρουσιακής ε, στάσης προς το Ιράν, ιδιαίτερα εάν το Κογκρέσο προχωρήσει σε κυρώσεις. Αλλά αυτό ενισχύει την σημασία όσο και την ευθύνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιζητήσει το διάλογο με το Ιράν και μεταξύ του Ιράν και ε, διαφόρων ε, δυνάμεων της περιοχής για να αποκλιμακωθεί και να ε, συγκρατηθεί η βία. Και τέλος, να πω δύο λόγια για την ιστορία του κυβερνοχώρου στη Μέση Ανατολή. Δεν πρωταγωνιστεί σήμερα στη σύγκρουση, αλλά μπορεί στο μέλλον να γίνει. Και αυτό θα πρέπει να το δούμε και στο ρωσικό πλαίσιο, γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Το έχουμε παραβλέψει. Τα τελευταία χρόνια, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, η Μέση Ανατολή έχει γίνει μέτωπο ε, γεωπολιτικών στον κυβερνοχώρο. Μπορεί να ξέρετε ότι το Ισραήλ για μια δεκαετία είναι μεγάλη δύναμη στο διαδικτύο, αλλά από το 2012 Ε, την επίθεση με ιό ε, σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις, Ισραήλ και ΙΠΑ, έχουν ε, απαντήσει το, Ιράν με επιθέσεις κυβερνοεπιθέσεις και οι χώρες της συνεργασίας, το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου προσπαθούν να προχωρήσουν και το τελευταίο επεισόδιο ήταν ο αποκλεισμός στο Κατάρ το καλοκαίρι το οποίο ξέρετε ότι μπορεί να προήλθε ε, από χακάρισμα ιστοσελίδας ε, του Κατάρ. Υπάρχουν κυβερνοεπιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Δεκαπλασιάστηκαν, για να μην πω δέκα, πενταπλασιάστηκαν την τελευταία πενταετία. Το Ιράν ταυτόχρονα είναι και το μεγαλύτερο θύμα αλλά και ο μεγαλύτερος θήτης των περίφημων ε, κρατικοδίαιτων επιθέσεων. Και είναι τώρα μια κόντρα αυτή, μια σύγκρουση μεταξύ των χωρών συνεργασίας του Περσικού κόλπου, ε, του Ισραήλ και του Ιράν. Είναι, σχεδόν, είναι εύκολο αυτό και φτηνό ε, να γίνει κυβερνοπόλεμος και εύκολο για το Ιράν. Είναι χαμηλός ο κίνδυνος αντιπίνων Δηλαδή έχει μεγάλο αντίκτυπο με χαμηλό κόστος και χαμηλό ρίσκο. Και αυτό είναι τμήμα της στρατηγικής της επεκτατικής του Ιράν που εξάγει τώρα στον κυβερνοχώρο ε, τον πόλεμο δια αντιπροσώπων. Χρησιμοποιεί ομάδες hacker αντίστοιχες με κίνηση της Ρωσίας. Το να χρησιμοποιήσει τώρα αντιπροσώπους και στον κυβερνοχώρο είναι ένας επιπλέον κίνδυνος. Πέρα από τη μεταφορά της τεχνολογίας, σε αντίθεση ε, με ε, τα συμβατικά όπλα, τα τεχνολογικά όπλα χρειάζονται νέα τροφοδοσία και επίσης δεν είναι και δεδομένη η αφοσίωση και η πίστη αυτό το hacker που μπορεί να αλλάξουν στρατόπεδο. Ε, και αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα νέο πυλώνα της στρατηγικής του Ιράν κάνουν έτσι αποτελεσματικές ενέργειες ε, που δεν θα μπορούσαν σε στρατιωτικό επίπεδο γιατί δεν έχουν τις δυνατότητες και τις ικανότητες. Και τώρα έρχεται η Σαουδική Αραβία ε, που είναι ευάλωτη. Γιατί υπολείπεται κατά πολύ στον κυβερνοχώρο η Σαουδική Αραβία σε σχέση με το Ιράν. Και το γεγονός ότι τα έχει κάνει τώρα πλακάκια με το Ισραήλ που είναι ε, ε, ε, η δύναμη στον κυβερνοχώρο δεν είναι τυχαίο και μπορεί να αντισταθεί στο Ιράν. Υπάρχουν κάποιες εντάσεις εκεί, οι οποίες επιταχύνονται με το ίντερνετ και εντείνονται ήδη φυστάμενες εντάσεις ακόμα περισσότερο στην περιοχή. Ευχαριστώ. So who was first? Mr. Killam? Mr. Carver's coordinator. Mm-hmm. Okay, so we start with the coordinator. Πρώτα-πρώτα η ερωτήση από πλευρά των συντονιστών. Κύριε Κάρβερ. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Ναρμπόνα. Μας ε, Είπατε για το κοσμικό κράτο που ξαπλώνεται στην Μέση Ανατολή, που διαδίδεται ας πούμε περισσότερο και τι με τις δυσκολίες στο Βόρειο Ιράκ, ε, στη Συρία, ε, όλοι αυτοί που ε, έχουν χτυπηθεί από την κατάσταση. Το Ισλαμικό κράτο που έχει συρρικνωθεί στο 5% όσον αφορά την κατοχή εδάφου. Και επίση είπατε για την παρουσία τζιχαντιστών στην ε, Αραβική Χερσόνησο. Για πέστε μας. Αναφέρατε το, ότι μπορεί να αποκτήσει κάποιο ρόλο η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, όσον αφορά τον πόλεμο στην Ιεμένη. Για εξηγήστε μας. Και πώς βλέπετε την ακεραιότητα, την εδαφική της ε, Ιεμένης. Είναι δυνατόν η Εμένη να μείνει ως έχει. τι θα γίνει και για τη Βόρεια και τη Νότια Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να επηρεάσει τη Σαουδική Αραβία όσον αφορά την πολιτική της. Και μήπως θα υπάρξει προστριβή σε σχέση με το Brexit, με τη ΣΥΠΑ, μεταξύ ΥΠΑ δηλαδή, και Ευρωπαϊκής Και εγώ θέλω το Brexit, αλλά πέστε μας πώς θα επηρεάσουν αυτές οι προστριβές ε, την εμπλοκή μας στο ΝΑΤΟ και έλα. Πολύ επίκαιρα αυτά που μας είπατε για την πληροφορική, και τα σχετικά προβλήματα. Ε, το θέμα αυτό είναι καυτό γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χάσει το τρένο. Έχει μείνει πολύ πίσω. Επίσης όσον αφορά την αντιπαράθεση στην Ιεμένη, εκπονούμε τώρα κάποιο σχετικό ψήφισμα. Θα πρέπει να ανοίξουν διάβλη για ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό θέλει το Κοινοβούλιο. βλέπουμε ότι πάει να κλείσει το ένα μέτωπο. Ε, δεν τέλειωσε ο πόλεμος, αλλά πάει να κλείσει. Αλλά βλέπουμε να ξανοίγονται καινούριες αντιπαραθέσεις. Με το Ιράν, το Ισραήλ. Για πέστε μας. Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι ομοιότητες μεταξύ των τρομοκρατών, Σουνιτών και Σίτων όλοι τους θέλουν να απαλλαγούν από οποιαδήποτε επιρροή της Δύσης. Να απαλλαγούν από τους Δυτικούς και το Ισραήλ. Ο ρόλος του Ιράν, τι λέτε. Έχουμε το ψήφισμα του Κοινοβουλίου και εκεί λέμε ότι το Ιράν θεωρούμε ότι είναι συμμαχός μας κατά της τρομοκρατίας. Όμως ε, θεωρήθηκε ότι είναι ο μεγαλύτερος εξαγωγής τρομοκρατών. Επίσης, είχαμε συνάντηση του Ρευγού Συνδέσμου σε επίπεδο πολλών εξωτερικών. Γι' αυτό. Εσείς πώς βλέπετε τον ρόλο της χώρας του Ιράν δηλαδή. Πολύ σημαντικό. Ε, γιατί τρέφαμε ελπίδες για τον ρόλο του Ιράν. Όμως είδατε ποια είναι η θέση του ε, ΝΥΠΑ και του Ραβικού Συνδέσμου. Χθες ο πρόεδρος Ασάντ πήγε στο Σότσι και συνάντησε τον πρόεδρο Πούτιν. Και τώρα θα συναντήσει Τούρκους και Ιρανούς ο Πούτιν. Και επίσης κανονίζεται συνάντηση στο Σότσι όλων των εμπλεκομένων στη, στο πόλεμο της Συρίας. Σκοπός είναι η πύλη των διαφορών και από ό,τι καταλαβαίνω η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να προχωρήσει η διαδικασία των Βρυξελών. Εσείς τι λέτε. Έχει πολιτικές και ηθικές ευθύνες ο πρόεδρος Άσαντ. Ανθρωπιστικά εγκλήματα. Έχουμε και εγκλήματα πολλά για τα οποία φέρει την ευθύνη. Ευχαριστώ. Φρόνιντ. Ευχαριστώ πολύ. Λυπάμαι που άργησα. Συγχωρήστε με, δεν μπορώ να σχολιάσω τα του κυρίου Ναρμπόνη, γιατί δεν ήμουν εδώ. Πάντως, να σας μιλήσω για κάτι που είπε η κυρία Κάους στην εισήγησή της. Θα σταθώ σε κάποια σημεία από όσα μας ανέφερα. Το πιο ενδιαφέρον είναι η αντιπαράθεση Ιράν και Σαουδικής Αραβίας. Φυσικά αρνητικά ενώ ότι παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι πηγή ανησυχία. Δεν διαμεσολαβεί καθόλου η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ανέκαθεν ήταν το πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουλάχιστον όσο εγώ ασχολούμαι τις πιο πρόσφατες δεκαετίες, μια που εκπροσωπούμε 500 εκατομμύρια. Είμαστε μία από τις ε, πιο ισχυρές οικονομίες παγκοσμίω. Παρ' όλα αυτά, μένουμε άπραγοι και να το πω διπλωματικά όσον αφορά αντίδραση ή παρέμβαση σε κάποια κρίση. Και μιλώ για κρίσεις που μας ε, θίγουν ή θα μας θίξουν. Το ίδιο ισχύει και όσον αφορά την αντιπαράθεση της Σαουδικής Αραβίας και Ιράν. Το πρόβλημα κατά τη γνώμη μου είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως σωστά είπατε, έχουν πάρει συγκεκριμένη τοποθέτηση υπέρ του Ισραήλ, και της Σαουδικής Αραβίας. Υπάρχει πρόβλημα με τη Σαουδική όχι τόσο με το Ιράν. Υπάρχουν καλύτερε σχέσει. Όμω. Αν εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτή την αντιπαράθεση Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, μάλλον θα βρεθεί αντιμέτωπη με τις Ηνωμένε Πολιτείες. Είμαστε σε αντίθεση με τη δική τους πολιτική. Ε, δεν το βλέπω αυτό. Δεν βλέπω να κοντράρουμε την σημερινή Αμερικανική κυβέρνηση. Άρα, τι λύση θα προτείνει για αυτό το πρόβλημα. Από τότε που έγινα ευρωβουλευτής, πάντοτε ήμουν υπέρ του να έχουμε πιο ισχυρή εξωτερική πολιτική και όχι μια πολιτική που επεμβαίνει εκ των υστέρων. Α, στη Συρία τίποτα δεν κάναμε. Α, και ο κύριος Κέλαμ μας τα εξήγησε. Μας είπε και για τη συνάντηση στο Σότσι. Απουσιάζει από το τοπίο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, με όλα αυτά όμως μας αφορούν πάρα πολύ που για να παρέλθω στο θέμα τη Σαουδική Αραβία και Ιράν, εσεί τι ρόλο βλέπετε ότι μπορεί να διαδραματίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση χωρί να κοντράρετε με τι Ηνωμένε Πολιτείε και έτσι να θέσουμε κινδύνο τις ε, διατλαντικές μας σχέσεις. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ. στα πολωνικά θα σας τα πω. Ευχαριστώ λοιπόν πολύ για τις παρουσιάσεις σας και την ανάλυση που μας παρουσιάσατε. Αυτό που ήταν πολύ ενδιαφέρον για μένα ήταν αυτό που είπε η κυρία Κάους. Κυρίως για τα διαρθρωτικά ζητήματα. Αυτή η διαρθρωτική δηλαδή σύγκρουση ανάμεσα στην Σαουδική Αραβία και το Ιράν και το ενδιαφέρον που δείχνει η διεθνή κοινότητα θα πρέπει να οδηγήσει στην αποφυγή πολέμου. Μας ενδιαφέρει η ασφάλεια γενικά και τρίτων χωρών και όχι μόνο στην περιοχή και αλλού. Αλλά όπως είπατε είναι διαρθρωτικό πρόβλημα. Δεν είναι δηλαδή μια διμερή σύγκρουση, αλλά έχει να κάνει με την πολιτική του Ιράν που έχει επεκτατικές τάσεις. Χρησιμοποιεί λοιπόν το Ιράν πυρηνικές συμφωνίες προκειμένου να μην βελτιώσει τελικά την οικονομική του κατάσταση, αλλά προκειμένου να νομιμοποιήσει τις επιθυμίες του για επέκταση στην περιοχή. Οπότε το πρόβλημα δεν είναι το πώς θα αποφύγουμε την ενίσχυση των εντάσεων μεταξύ δύο ομάδων χωρών, αλλά πώς θα αποφύγουμε η πολιτική του Ιράν να οδηγήσει σε τραγικές καταστάσεις. Ποια θα ήταν η αναλλακτική λύση να στηρίξουμε χώρες που θα μπορούσαν να σταματήσουν τις φιλοδοξίες του Ιράν, για παράδειγμα. Όταν μιλάμε για τις δραστηριότητε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, νομίζω ότι στην περίοδο κυρίως πριν αρχίσει ο στη Συρία και πριν αναμειχθεί η Ρωσία, φαίνεται ότι η κύρια φιλοδοξία του Ασάντ ήταν να διατηρηθεί στην εξουσία. Και τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή να καθίσουμε και να σκεφτούμε πώς θα αποσύραμε την στρατιωτική δύναμη της Συρίας στο Λίβανο. Το Ιράν δεν αγωνίζεται για επιβίωση, αγωνίζεται για να επεκταθεί και είναι έτοιμο να φτάσει σε ακραία μέσα γι' αυτό. Βλέπετε πώς συμπεριφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης της συμφωνίας ανέβαλα τα προβλήματα, δεν τα έλυναν. Οπότε τι θα μπορούσε να λειτουργήσει καλύτερα για να σταματήσουμε αυτή την επεκτατική διάθεση του Ιράν, τι θα μπορούσαν να κάνουν οι χώρες που είναι κατά αυτού. Ε, θέλετε συμπληρωματική ερώτηση εσείς παρακαλώ. Ναι, ναι. Αυτά που είπατε για τον ε, ρόλο μας στη Ιεμένη και πώς ε, αυτό θα μπορούσε να παρέμβει στο σχέδιο δράσης, το JCPOA. Και εγώ ήθελα τον λόγο, λέει πρόεδρος. Μιλάω τώρα όχι ως πρόεδρος, αλλά ως μέλος της Επιτροπής αυτής και έχω να κάνω και εγώ κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, αυτά που ακούσαμε για το ρόλο του Ιράν που είπε ο κύριο Ναρμπόνε και μετά αυτά που είπε η κυρία Κάτσο επίση για τον κυβερνοχώρο. Ρωτάω λοιπόν. Εδώ δεν είναι θέμα ευθυγραμμισμού του Ιράν με τη Ρωσία, δηλαδή δεν εμπίπτει στα σχέδια τα πολιτικά της Ρωσίας για τον κυβερνοχώρο. Για καιρό ανέπτυξαν τις δραστηριότητε τους σε αυτό το κλάδο. Μήπως δηλαδή τελικά αυτή είναι η μεγάλη απειλή. Και από τη Σαουδική Αραβία. Βέβαια το Ισραήλ έχει τέτοια μεγάλη δύναμη εδώ και καιρό. Και το Ιράν τώρα, όπως είπε ο κύριος Ναρμπόνε πολύ σωστά, παίζει περίεργο ρόλο στην περιοχή, όχι τόσο θετικό. Έχουμε εικόνες του στρατηγού Σουλεϊμάνη, για παράδειγμα, χτες ή προχτές, στη Συρία, που ανακοίνωσε το τέλος του ISIS, του λεγόμενου Ισλαμικού κράτους, το οποίο όμως βρίσκεται αλλού, έτσι, χωρίς ε, θετικά αποτελέσματα. Θα ήθελα λοιπόν να ακούσω και τους δυο σας να σχολιάσετε το ρόλο της Ρωσίας. Εκτός από τη συνάντηση στο Σότσι, γενικά Πώς βλέπετε εσείς τον ρόλο της Ρωσίας. Ακούσαμε για τις Ηνωμένε Πολιτείε, για την κυβέρνηση Τραμπ και μερικές φορές δεν πρόκειται μόνο για το λευκό οίκο, πρόκειται και για κάτι ευρύτερο. Και εμείς ε, σε αποστολή που είχαμε στι Ηνωμένε Πολιτείε, ακούσαμε μια καλή ισορροπία απόψεων. Και θα έλεγα ότι δεν είναι και τόσο υπέρ. Οπότε την αντίληψη αυτή για τις Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τη δούμε ευρύτερα και να λάβουμε υπόψη μας περισσότερους παράγοντες. Φυσικά και όλους μας απασχολεί η κατάσταση στην Ιεμένη. Συμμερίζομαι αυτά που λέει ο κύριος Κέλλαμ. Ότι δηλαδή πρέπει να κάνουμε έκκληση να ανοίξουν οι ανθρωπιστικοί οδοί προς τη χώρα αυτή. Αλλά πρέπει να θυμίσω την κατάσταση πριν από μερικά χρόνια, τότε που όλοι μας και με την συμμετοχή χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης θέλαμε να πιέσουμε αυτή τη χώρα που είναι μια από τις στοχότερες του κόσμου σε αυστηρές οικονομικές μεταρρυθμίσεις που ήταν πολύ δύσκολες για την κοινωνία την Ιεμενική και ίσως αυτό άνοιξε το δρόμο στη συνέχεια στη χρήση διαφόρων τεχνικών εκεί και με τη βοήθεια του Ιράν, φοβάμαι. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω κυρίως την κυρία Κάους για τις επιπτώσεις στη μετανάστευση της κατάστασης ε, της σύγκρουσης στην Ιεμένη. Όταν έχουμε βομβαρδισμούς στη Συρία, φυσικά υπάρχουν κύματα ε, μεταναστευτικά. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι και ο Σάντ έχει κάποια σχέδια για να διώξει ο πληθυσμό από εκεί. και πού πάνε οι άνθρωποι από την Ιεμένη, οι μετανάστες, ποιος τους παίρνει, πού βρίσκονται, ποια είναι η τύχη τους. Οπότε θα σας δώσω το λόγο με την ίδια σειρά. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ευρυφάσμα ερωτήσεων και θα προσπαθήσω να τις συγκεντρώσω κάπως για να τις απαντήσω. Αρχίζω με το ρόλο του Ιράν και με το τι μπορούμε να κάνουμε ώστε να μειώσουμε τις περιφερειακές δραστηριότητες του Ιράν, τις επεκτατικές. Προφανώς το Ιράν αναμειγνύεται και άμεσα και έμεσα σε διάφορα πεδία. Η ανάλυση μπορεί να διαφέρει για το ποιος είναι ο απευθείας ρόλος του Ιράν στην Ιεμένη αλλά αυτό που είναι προφανές είναι ότι το ΡΑΝ παίζει κάποιο ρόλο. Βέβαια το ερώτημα που τίθεται στη συνέχεια είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση τα γνωρίζει όλα αυτά. Και έρχονται προς συζήτηση στις επαφές που έχουμε με το Ιράν. Το κύριο ζήτημα είναι ότι διαφοροποιούμαστε όσον αφορά την προσέγγιση μας. Η Πυρηνική Συμφωνία για την Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει. Είναι κάτι πολύ σημαντικό διπλωματικά για τη μη διάδοση των πυρηνικών. Είναι σημαντικό βέβαια στη στρατηγική μας να χωρίζουμε τα πράγματα. Όπως είπα, υπάρχουν ανησυχίες για το Ιράν, το οποίο εμπλέκεται έμεσα σε συγκρούσεις με εμπόλεμες ομάδες. Αλλά αυτό πρέπει να μείνει διακριτό στο διάλογό μας με το Ιράν γιατί υπάρχει και η πίεση της απομόνωσης. Οπότε ο ρόλος που μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι να του δείξει ότι δεν θα βρεθεί και πάλι στην απομόνωση. Στην Ιεμένη είπα ότι φαίνεται πως η διπλωματία δεν αποφέρει καρπούς. Υπάρχει κλιμάκωση, περισσότερες εντάσεις. Συγχρόνως όμως είναι αλήθεια ότι αντιλαμβανόμαστε ότι ο πόλεμος δεν ε, πέτυχε αυτά που θέλαμε, παραμένει αστάθεια, ανθρωπιστική βοήθεια χρειάζεται, η πίεση προς την Σεουδική Αραβία ενισχύεται, επηρεάζει την πολιτική της Σεουδικής Αραβίας το γεγονός ότι δεν μπορεί να κερδίσει αυτή τη σύγκρουση κάτι το οποίο οδηγεί με τη σειρά του σε άλλους παραγόντες αστάθειας. Ενίσχυση τρομοκρατικών ομάδων, για παράδειγμα. Ε, στρατιωτική κλιμάκωση. Όλα αυτά τα στοιχεία παίζουν ρόλο. Και νομίζω ότι πρέπει να τα λάβουμε υπόψη μας στο διάλογό μας με τη Σαουδική Αραβία και άλλες χώρες του κόλπου. όλα τα ζητήματα πρέπει να μπουν στο ευρύτερο πλαίσιο της περιοχής, γιατί στο κάτω-κάτω στην περιοχή του κόλπου είμαστε σε μια κατάσταση όπου συνεχίζουμε να βλέπουμε να κλιμακώνονται οι πιέσεις. Πώς βλέπουμε τις απειλές, ποια είναι η πραγματικότητα των απειλών και πολιτικά και αλλιώς όλα αυτά τα στοιχεία επιδεινώνουν την κρίση και τη, ενισχύουν τις ε, εντάσεις. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας τη μεγάλη εικόνα στην περιοχή και να προσπαθήσουμε να βρούμε τρόπους αποκλιμάκωσης με τη συμμετοχή όλων των πλευρών, με πίεση, με διάλογο και μόχλευση. Στη Συρία, για παράδειγμα. Βέβαια στη Συρία είναι κυρίως στρατιωτικοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Η Ρωσία σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρουμε όμως ότι ακόμα και αυτοί που έχουν στρατιωτικό ρόλο έχουν τη δική τους πίεση. Η Ρωσία σίγουρα προσπαθεί να χρησιμοποιήσει τη νίκη της, αλλά έχει και ανησυχίες να μην παγιδευτεί και να δει τι θα γίνει μετά με την ανοικοδόμηση. Γενικά κοιτάει τα πιο μακρινά συμφέροντα. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι το οποίο μπορεί να λειτουργήσει ως μόχλευση για την κατάσταση μετά την σύγκρουση στην περιοχή και για την ανοικοδόμηση. Δηλαδή, αυτό που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει είναι να ακολουθήσουμε τη λογική της αποκλιμάκωσης. Και αυτό εννοούσα. Αυτό είναι ένα χείρημα που δεν μπορεί κανείς να το κάνει από μόνος του, στη γωνιά του. η Ευρωπαϊκή Ένωση ήδη χρησιμοποιεί ό,τι μέσα έχει στη διάθεσή της προκειμένου να βάλει όλες τις πλευρές να βοηθήσουν με προβληματισμούς. Ας πούμε, ποιο είναι το μέλλον της τρομοκρατίας, κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Φυσικά υπάρχουν διαφορετικές ομάδες που βασίζονται στη λογική του κατακαιρματισμού αλλά τελικά είναι προς το συμφέρον όλων των πλευρών να απαλείψουμε την τρομοκρατία. Να λοιπόν ένας τομέα συνεργασίας που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ώστε να μπούμε και στη διαδικασία αποκλιμάκωσης. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα κυρία Κάους, παρακαλώ. Thank you. Ευχαριστώ. Ωραία. Από πού να αρχίσω. Από τον κύριο Φρόιντ. Σημαίνει κόντρα με τις Ηνωμένε Πολιτείε αν αναμειχθούμε ε, στη σύγκρουση ε, Ιράν-Σαουδικής ε, Αραβίας. Οι Ηνωμένε Πολιτείε όταν λέτε τι ακριβώς εννοείτε Ποιου ακριβώ εννοείται. Γιατί δεν <coughs> μιλούν με μία φωνή αυτό τον καιρό. Και θα πρέπει να ξεφύγουμε από τη λογική αυτή που έχουμε ότι μιλάμε μόνο με την πρώτη ή τη δεύτερη γραμμή της κυβέρνησης. Υπάρχουν εξέχουσες προσωπικότητες που στο Κογκρέσο ας πούμε και ρεπουμπλικανοί εξέχονται συμφωνούν με την ευρωπαϊκή θέση για το Ιράν. Υπάρχει πολύ περιθώριο για άσκηση πίεσης, ιδιαίτερα στο Κογκρέσο αυτές τις κρίτιμες ε, εβδομάδες. Ξέρω ότι έχουν εμφανιστεί απεσταλμένοι ε, από την Ευρώπη, Γερμανία, Γαλλία, Βρετανία, ε, στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο, στο Κογκρέσο, για να διασπείρουν πούμε, τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κατά τα άλλα δεν νομίζω ειλικρινά να υπάρχει πρόβλημα να διαφωνήσουμε ε, με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Σε πολλά σημεία διαφωνούν οι Ηνωμένε Πολιτείε με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν το βρίσκουν και μέγα πρόβλημα. Ε, ε, I don't think δεν νομίζω λοιπόν ότι αυτό συνιστά σύγκρουση. Βεβαίως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διευρύνει την επικοινωνία της με το Ιράν που έχει ε, πλεονέκτημα και ως προς το ύφος της επικοινωνίας και ως προς τους διάβλους που έχουμε. Αλλά δεν νομίζω η Ευρωπαϊκή Ένωση να πρέπει να είναι διαμεσολαβητής μεταξύ Ιράν και Σαουδικής Αραβίας, απλώς να πιέσει τις Ηνωμένε Πολιτείες, όπως είπα προηγουμένως η συμπεριφορά της Σαουδικής Αραβίας δεν θα ήταν τέτοια σήμερα αν δεν του στήριζαν οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εν Και μην ξεχνάμε ότι ορισμένοι παράγοντες εκεί δεν θέλουν αποκλιμάκωση. Κλιμάκωση θέλουν και το Ιράν και εν μέρει η Σαουδική Αραβία. and in Lebanon, Israel. So, um... Και στο Λίβανο και στο Ισραήλ. Ας μην υποθέτουμε ότι όλοι θέλουν αποκλιμάκωση και θα έρθει ως εκθαύματος γιατί κανείς δεν επιθυμεί τη σύγκρουση. Ίσα ίσα είναι πολλοί εκείνοι που πιέζουν για τη σύγκρουση. Για το Ιράν βεβαίως είναι διαρθωτικό το πρόβλημα και κανείς δεν τρέφει εδώ αυταπάτες ως προς την περιφερειακή πολιτική της, ε, του Ιράν. Είναι ε, άκρος ε, κατασταλτική και επεκτατική και τα σχέδιά τους τα γνωρίζουμε. Αλλά τι θα κάνουμε εμείς. Μέχρι τώρα η Σαουδική Αραβία ποτέ δεν προσπάθησε σοβαρά να αρχίσει διαρθωμένο διάλογο με το Ιράν. Αυτό μπορεί να γίνει διμερός ή περιφερειακά με κάποιους παράγοντες, αλλά όχι ε, με μεσάζοντα τις ΗΠΑ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν θα πρέπει εμείς να ασκήσουμε την πίεση που μπορούμε με τους μοχλούς που έχουμε. Δεν το έχει προσπαθήσει αυτό η Σαουδική Αραβία και είναι και προς το δικό της συμφέρον. Δεν έχει νόημα να συνεχίσει αυτή την τακτική. Έχει και αρνητικές επιπτώσεις για την ίδια. Τι άλλο τώρα. Σε σχέση με αυτό που είπατε εσείς, Πρόεδρε, για το ρόλο της Ρωσίας ε, και τον κυβερνό πόλεμο. Αυτό σημαίνει ότι έχει ευθυγραμμιστεί το Ιράν με τη Ρωσία. Εγώ δεν θα το πήγαινα μέχρι εκεί. Δεν ξέρω. Τι ανταλλαγές γίνονται μεταξύ Τεχεράνης και Μόσχας. Ε, μπορεί να έχουν διδαχθεί από τη Ρωσία μερικά πράγματα, δεν σημαίνει ότι έχουν ευθυγραμμιστεί κιόλα. Και για να είμαι ειλικρινή, οποιοδήποτε στον κόσμο που παρατήρησε την επιρροή που έχει η Ρωσία στις εκλογές στην Ευρώπη και στις Ηνωμένε Πολιτείες τα τελευταία χρόνια, και οποιοδήποτε έχει επεκτατικές βλέψεις μπορεί να διδαχτεί παρατηρώντας αυτά. Ε, δεν είναι μυστικά, ούτε χρειάζονται μυστικές επικοινωνίες και πληροφορίες. Ε, σε κάποιο βαθμό συγκλίνουν με τη Ρωσία και αλλού διαφωνούν. Δεν σημαίνει ότι ευθυγραμμίζεται πλήρως το Ιράν. Γενικά όμως, η επιστροφή της Ρωσίας στη Μέση Ανατολή είχε και αυτό το στοιχείο. Μεταξύ άλλων. Έχω την αίσθηση ότι ενδιαφέρεται λιγότερο για τη Μέση Ανατολή και περισσότερο για τον Ασάντ και να κερδίσει ε, σημασία ε, σε μια περιοχή που είναι κομβική σημασία για έναν από τους ε, αντιπάλους της. Δηλαδή, όσο περισσότερο συγκρούεται το Ιράν με τις ΗΠΑ, τόσο σημαντικότερο θα είναι και για την ίδια τη Ρωσία κατά κάποιο τρόπο. Η εμένη μετανάστευση. Δεν έχω αριθμητικά στοιχεία. Αυτό το δίνουν ε, ε, οι υπηρεσίες του ΙΕ που ασχολούνται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Αλλά οι μετανάστες που θα πάνε για να φύγουν από εκεί δεν θα πάνε στο Ρωμάν, στη Σαουδική Αραβία θα πάνε. Τι άλλο, τι άλλο. Κύριε Κέλαμ, Χαίρομαι πολύ που άκουσα για το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ελπίζω να μην μείνει κάπου μετέωρο, αλλά να οδηγήσει και σε κάποια δράση. Ρωτήσατε ε, για τους εξτρεμιστές αν υπάρχουν ομοιότητες μεταξύ Σουνιτών και Σιητών. Δεν ξέρω αν κατάλαβα τι εννοείται ακριβώς. Ποιους εξτρεμιστές. The different, uh, religious or identity... Υπάρχουν διαφορετικοί διάφοροι εξτρεμιστές με βάση τη σκεφτική ιδεολογία στη Μέση Ανατολή. Είναι μια ιδεολογία που δικαιολογεί, ε, αλλά εξυπηρετεί πολιτικές σκοπιμότητες. Οπότε δεν έχει νόημα αν, έχει, αν είσαι εκεί Σιήτης ή Σουνίτης. Δεν ξέρω αν θέλετε να το συζητήσουμε, να το συγκεκριμενοποιήσετε περισσότερο για να σας απαντήσω. Συνάδελφοι, μπορείτε να συνεχίσετε τη συζήτηση, αλλά... Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο και έχουμε και άλλο θέμα στην ημερήσια διάταξη μέχρι τις 12.30. Προτείνω να το αναβάλουμε αυτό για την επόμενη συνεδρίαση. Θα παρακολουθούμε την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Συνεχώς ε, και αδιαλείπτως. Είναι τόσο σημαντική και τόσο δυναμική στις εξελίξεις και για θέματα ασφαλείας πάντα μας απασχολούν αυτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε. Ας τους χειροκροτήσουμε. Μην Μη φύγετε, έχουμε και άλλο θέμα. Και λιγότερο από 20 λεπτά για την ενημέρωση της αποστολής ΕΝΤΕ ΑΦΕΤ στην Ουάσιγκτον και το Νόρφολκ, Βιρτζίνια. Uh, τα έγγραφα αυτά θα έχετε που αφορούν αυτή την κοινή αποστολή. Προεδρεύουσα στις υποφαινόμενες αλλά και συμποδέμου του κύριου Μακάλιστερ. Πήγαμε στην Ουάσιγκτον ε, και στο Νόρφοκ της Βιρτζίνια. Ε, για να επισκεφτούμε το στρατηγείο SACT που βρίσκεται εκεί στην Βιρτζίνια στο Νόρφοκ. Οπότε το έτοιμά μας ικανοποιήθηκε και κάποια στιγμή η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε να γίνει κοινή η αποστολή με την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων Εγώ είπαμε να προεδρεύσω στις επαφές μας του ΝΑΤΟ στο Νόρφοκ και ο Ντέιβιντ Μακάλιστα προεδρεύσε στις περισσότερες αντίσεις στην Ουάσινγκτον εκτός από την ανταλλαγή απόψεων με κάποιους ε, ειδικού από το Ατλαντικό Συμβούλιο αυτά σε κάποιο δείπνο εργασία. Ήταν μια εκδήλωση πολύ ενδιαφέρουσα. Η αποστολή ξεκίνησε 31 Δεκάτου και διήρκεσε μέχρι τις 3 ε, Νοεμβρίου την ε, πρώτη μέρα. Είχαμε την άφηξη το απόγευμα και το βασικό μας θέμα ήταν ε, μια ενημέρωση από αυτά γίνανε στην πρεσβευτική κατοικία. Ο πρέσβης, ο κύριος ο Σάριβαν, επικεφαλής αντιπροσωπείας μας. Μας ενημέρωσε για την περίπλοκη κατάσταση όσον αφορά ε, τα πολιτικά και τις εξελίξεις στην ε, Αμερική και βέβαια Συζητήσαμε για τα τη συμφωνίας με το Ιράν, από πυρηνικοποίηση, συζητήσαμε τα πιθανά σενάρια. Και αυτά, λίγο αφού ο πρόεδρος Τραμπ είχε προβεί στην ε, ανακοίνωση να αρνηθεί να αποπιστοποιήσει την συμφωνία Οπότε και είχαμε την παρουσίαση των σενάριων που σας ανέφερα πλευράς του πρεσβευτή, του κ. Σάλιβαν. Συζητήσαμε τις σχέσεις με ΝΑΤΟ και Ηνωμένες Πολιτείες, τις διατλαντικές, υπερατλαντικές πολιτικές μας. Πρόκειται για παραδοσιακές σχέσεις μας επί πολλές περιόδους ε, διακυβέρνηση από διαφορετικές κυβερνήσεις της Αμερική συζητήσαμε μετά της παγκοσμίου ασφαλείας και μετά στο Νόρφοκ της ε, Βιρτζίνια για να φτάσουμε εκεί βέβαια το ταξίδι κράτησε πολλή ώρα. Όμως η γραμματεία μας και μπράβο τους κατάφεραν πάρα πολύ καλά να τα οργανώσουν τα του ταξιδιού αυτού. Μας φιλοξένησε εκεί το, το επιτελείο του ΝΑΤΟ επικεφαλής ήταν ο στρατηγός Μερσιέ, αλλά είχαμε τον Αβραχό Νίλσον, τον πτέραρχο Στέισι και τους διάφορους επιτελάρχες. Και συναντηθήκαμε ο κ. Μακαλιστέρ και υποφαινομένη με όλους τους, όλα τα κορυφαία στελέχη του, του, του επιτελείου και είχαμε πολύ ολοκληρωμένη ενημέρωση συζήτησαμε για τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα της κοινή ε, δήλωσης διακήρυξης της Βαρσοβίας Πολύ πολύ ενδιαφέροντα κάτι γνώμη μου. Και αυτά μόλις δύο-τρεις μέρες πριν την στρατηγική ανάλυση του ΝΑΤΟ. Μακρά συζήτηση όσον αφορά τις ε, απειλές και επικαιροποίηση των αναλύσεων και είχαμε και ένα γεύμα εργασία. Οπότε χωριστήκαμε σε μικρότερες ομάδες, να μιλήσουμε σε διάφορους αξιωματικούς. Σε υπαλλήλους από διαφορές χώρες. Σκεφτήκαμε και κάποιο πολεμικό σκάφος. Πώς λέγεται τόσο να το ξέχασα. Εκεί μας υποδέχθηκε βέβαια το πλήρωμα κυβερνήτης. Εξήγησαν τα, των αποστολών τους, τις διαδικασίες που ισχύουν Την ίδια μέρα επιστρέψαμε στην Washington. Και άρχισε η δουλειά πρωί-πρωί. Σαντίσαμε κάποιους ε, βουλευτές και από τα δύο μεγάλα κόμματα. Μίλησαμε με την ομάδα των βουλευτών που ενδιαφέρονται για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις. προείδρευσε από πλασά Αμερικανών ο κύριος Βίλσον πλευράς Ρεπομπλικάνων και ο Γκρέγορη Μίξ από πλευράς των ε, Δημοκρατών. Στη συνέχεια. Συναντήσαμε έναν ε, διευθυντή, έναν υψηλό βαθμό υπάλληλο του Υπουργείου Εθνικής Αμήνης του Πενταγώνου. Και εκεί έγινε μια πλήρης ενημέρωση για την πολιτική εθνικής αμήνης και στήσαμε τις ε, εξελίξεις στην Ευρώπη. Τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από πλευράς Ένωσης όσον αφορά την άμυνα και ασφάλεια. Κατά την ε, μεσημερινή διακοπή με τον David Μακάλιστερ συναντηθήκαμε με τον σύμβουλο α, ε, σύμβουλο του Αντιπροέδρου των Μανοπολτιών τον κύριο Οχάρα, τον στρατηγό Οχάρα επίσης, που είχε αντικαταστήσει την κυρία Τόμσον, που προήχθη κάπου στο Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ ενδιαφέρουσα και αυτή η συνάντηση. Το βασικό θέμα αφορούσε την κατάσταση στο Ιράν και διάφορα προβλήματα. Συζητήσαμε για τη Ρωσία, τη Μέση Ανατολή. Ε, φυσικά συζητήσαμε και για τα θέματα από του Ιράν συνολικά την πολιτική μας ως προς το Ιράν οπότε και η πλειοψηφία των ε, συναδέλφων ξεκάθαρα ε, τοποθετήθηκαν γι' αυτό και για άλλα ζητήματα όσον αφορά τον ρόλο του Ιράν στην ευρύτερη περιοχή όσον αφορά την χρηματοδότηση του Ιράν προς τρομοκράτες. Συζητήσαμε τα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και πιο συγκεκριμένα συζητήσαμε για τη σειρά εκτελέσεων που, έχουν, που είχαν προηγηθεί για την καταδίκη ανηλίκων και νέων γενικά θέματα δηλαδή εκτός του πυρηνικού μήνυμα που στείλαμε είναι το ότι οι εξελίξει του Ιράν απασχολούν σοβαρά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι μας απασχολεί το ότι αποσύρεται από τη συμφωνία ε, η χώρα, οι Ηνωμένες Πολιτείες. και σε περαιτέρω συναντήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίστηκε ότι οι εξελίξεις έχουν να κάνουν με κάποιες εσωτερικές εξελίξεις και κάποιες επιλήψιμες διαδικασίες και εξελίξεις σε σχέση με την συμφωνία, τη σύναψη αυτής. Και πολλοί από τους αγορητές είπαν ότι δεν θεωρούν ότι βρίσκεται κινδύνο ε, η συμφωνία και ότι θα συζητηθεί η υπόθεση στο Κόγκρεσο. Αργότερα έγινε κάποια κοινή συνάντηση στο Λευκό Οίκο με ε, τον Διευθυντή Εθνικής Ασφαλείας με τον Σύμβουλο Ευρωπαϊκών Θεμάτων και εκεί έγινε μια σύντομη αναφορά σε διάφορα ζητήματα. ό,τι θυμάμαι είχαμε την μακρά ζήτηση στο Ατλαντικό Συμβούλιο με τους εκπροσώπους των διαφόρων think tanks για σημαντικά ζητήματα ασφάλειας και άμυνας. και ο Φράντσις Μπράνουελ, ανώτερος, ανώτερος τέλεχος της Ένωση ε, Ένωσης, ε, προείδρευσε και είχαμε επίσης συμμετοχή ε, πάρει ψηλοβάθμων στελεχών και τον αναπληρωτή Υπουργό Εξωτερικών αλλά και τον αναπληρωτή Γενικό Νοματία του ΝΑΤΟ τον κύριο Ράσμπολ, πρέσβης και η επομένη ήταν η τελευταία μέρα της ε, εκεί διαμονής μας και ασχοληθήκαμε με κάποια πλήρη ενημέρωση από ανωτέρους ε, υπαλλήλου του Υπουργείου Εξωτερικών. Είχαμε δύο υφυπουργούς, μας ενημέρωσαν για συγκεκριμένα θέματα, δηλαδή για το Ιράν, για τις διαπραγματεύσεις με τη μη διάδοση των πυρηνικών, για θέματα ασφαλείας. Ήταν και κάποιος ε, επικεφαλής διαπραγματευτής με, την Κορέα, ως, επίσης συζητήσαμε αντιτρομοκρατική πολιτική και τη γενικότερη κατάσταση στην ε, Μεσανατολή και Βόρεια Αφρική. Από ό,τι θυμάμαι, αυτά. Έχετε το λόγο και παρακολουθεί να είστε σύντομοι. Όποιο θέλει. Κανεί. Καλά. καλά. Σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν. Θα ήθελα να σας θυμίσω ότι θα αρχίσουμε στις 2.30 στη συνέχεια. Μην το ξεχάσετε παρακαλώ στις 2.30 με τη δημόσια ακρόαση με θέμα η διάσταση της ασφάλειας της αλλαγής του κλίματος. Ποιες είναι οι επιπτώσεις. Σας ευχαριστώ.